Σαν, are you ready to start so we could start the meeting? Είστε έτοιμοι αγαπητοί συνάδελφοι να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα παρακαλώ να αρχίσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Το σημείο το πρώτο είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Σον Κέλλη για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές Ευρωπαϊκής Ένωσης του Διεθνές Ταμείου για την Ιρλανδία. Το λόγο έχει ο κύριος Σον ε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Το διεθνέ Ταμείο για την Ευλαβία λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γεννήθηκε μετά από την Αγγλοαβλιανδική Συμφωνία εδώ και 20 περίπου χρόνια. Η χρηματοδότηση ξεκίνησε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά. Το πρώτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε αυτή τη φάση μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ πάρα πολλοί πιστεύουν στην Ιρλανδία και πίστευαν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν αποκλειστικά υπεύθυνε για τη χρηματοδότηση του Ταμείου αυτού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βελτιωθεί η μορφή επικοινωνία μα προ τον Ιρλανδικό λαό και να πούμε το μεγάλο ποσοστό του ταμείου που προέρχεται από την Ένωση. Η νομική βάση ισχύει αναδρομικά από το 2007 και μετά. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάστηκε να περάσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αποκατασταθεί το νομικό πλαίσιο. και γι' αυτό παρέπεμψε το Συμβούλιο και την Επιτροπή ε, στο δικαστήριο. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Έχω έναν συνάδελφο εδώ από την Ιρλανδία που ήταν μέλος της κυβέρνησης από την περιοχή τη Μεθοριακή και μπορεί να σας βεβαιώσει ότι το ταμείο αυτό είχε τεράστια ωφέλη στα πλαίσια της προσπάθειας οικοδόμησης μέτρων ειρηνικών και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκε και ο αθλητισμός για να προωθηθεί η συνεργασία ανάμεσα στις κοινότητες. Υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης αυτών των μέσων. Πάντως, μέσω της πρώτης ανάγνωσης, μέσω του καθορισμού της νομικής βάσης θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ Σον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω <clears throat> τον Κέλλη για τη συμμετοχή του σε αυτή τη συζήτηση. Πράγματι εκατομμύρια έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα και η διαδικασία αυτή έχει σαν στόχο να αποκαταστήσει την, τον τακτό χαρακτήρα θα έλεγα της λειτουργίας του Ταμείου. Ιδρύθηκε το Ταμείο αυτό το 1986 από την Ιρλανδική και τη Βρετανική κυβέρνηση με στόχο την οικονομική και ε, κοινωνική πρόοδο στη Βόρεια Ιρλανδία και να μην υπάρχουν διακρίσεις για την ενίσχυση των περιοχών και από τις δύο πλευρές της Μεθορίου. Τώρα οι περισσότεροι από εμά δεν θυμόμαστε μια τόσο, περίοδο, τόσο μεγάλη περίοδο ειρήνης. Έχει παίξει λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία έχει παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία, έχει βοηθήσει τις κοινότητες και από τις δύο πλευρές της Μεθορίου και από τις δύο πλευρές των πολιτικών σχηματισμών της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο κανονισμός αυτός έχει μεγάλη σημασία λοιπόν. Έχει σημασία να ασχοληθούμε και με τη νομική βάση για το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία. Έχει μεγάλη σημασία να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατόν, προσδίδοντας νομική βεβαιότητα στους χρήστες του. Αυτό που θα ήθελα επίσης να κάνω εδώ, σαν μέλος το οποίο εκπροσωπεί πέντε από τις κομιτείες του νοτίου, των νοτίων συνόρων ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και το ΕΙΡΕ, είναι ότι δεν πρέπει να δίδεται η εντύπωση ότι μιλάμε για ένα νέο ταμείο, απλά προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες οβούσαν και εμείς θα ενισχύσουμε την έκθεση του Σον Κέλλη και θα την υπερψηφίσουμε. Είναι μια ευκαιρία εδώ για να ευχαριστήσω συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες που έχουν συνεισφέρει όλα αυτά τα χρόνια στο Διεθνές Ταμείο, είπα δηλαδή Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Η <clears throat> το η συνεισφορά του στη διεθνή αυτή προσπάθεια. Στο τέλος του 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της έχει δώσει κάτι λιγότερο από 305 εκατομμύρια ευρώ. Έχει υποστηρίξει πολλούς τομείς το Ταμείο αυτό, κατοικία, εκπαίδευση, αστυνόμευση, κοινωνική οργάνωση και ο Σον Κέλλη αναφέρθηκε και στον αθλητισμό. Δυστυχώς, σχετικά με την Ευρώπη και τις δωρήτριες χώρες αναφέρομαι, το Ταμείο αυτό έχει αρχίσει και φθήνει σε επίπεδο οικονομικών υποχρεώσεων αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, να δίνουμε στίγματα ελπίδας σε αυτούς οι οποίοι ωφελούνται από το Ταμείο αυτό και θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες από τις υπεύθυνε κυβερνήσεις έτσι ώστε να παραταθεί η χρονική ισχύ του Ταμείου αυτού. Οι δωρήτριες χώρες μπορεί να συνεχίσουν λοιπόν να δίδουν χρήματα. Ελπίζω να κακοφορήσουν οι διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται ανάμεσα στην Ιρλανδική και την Αγγλική κυβέρνηση. Από το 2007 μέχρι το 2013 στα πλαίσια του τρίτου προγράμματος ειρήνευσης ε, τρία δις προβλέπονται έτσι ώστε να ενισχυθούν μέτρα εμπιστοσύνης και στις δύο πλευρές της Μεθορίου. Ήμουν μέλος αυτού εδώ του Κοινοβουλίου όταν η κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε πριν από χρόνια. Το απόγευμα εκείνης της μέρας ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζακ Ντελόρ, ανταποκρίθηκε άμεσα και θετικά σε μια έκκληση η οποία ακολούθησε την κατάπαυση του πυρός και είπε ότι η Ευρώπη θα ανταποκριθεί με πολύ πρακτικό τρόπο. Πώς θα το κάνει αυτό. Υπήρχε η δυνατότητα μέσω του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία έτσι το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αύξησαν την χρηματοδότηση του Ταμείου αυτού και όχι μόνο, αλλά ξεκίνησαν και μια νέα πρωτοβουλία. Ήταν η πρωτοβουλία για το Ταμείο ε, Ανοικοδόμησης, Συμφιλίωσης και Ειρήνευσης για να καλυφθούν οι ανάγκες των κοινοτήτων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Η διαφορά ανάμεσα στο Ταμείο αυτό και το Interreg το περιφερειακό το οποίο είναι σημαντικό και αυτό για την περιοχή αυτή είναι ότι υπήρξαν επιπλέον πιστώσεις. Δεν αντικαταστάθηκαν οι πιστώσεις του Interreg από κάποια άλλα. Το πρόγραμμα Interreg λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει φτάσει τα 256 εκατομμύρια στην περίοδο 2007 μέχρι το 2013, προβλέπεται να φτάσει. Όπως σας είπα προέρχομαι από μια κομιτεία της περιοχής, είναι το Ντόνεγκαλ, είναι η Αλάσκα της Ιρλανδίας το Ντόνεγκαλ, από τη μία συνορεύει με τη Βόρεια Ιρλανδία και από την άλλη με τον Νότιο Ατλαντικό. Εμπλέκομαι στην εθνική πολιτική ζωή από το 1981 και κάθε φορά που πήγαινα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περνούσα από τη Βόρεια Ιρλανδία και εκτιμώ τους καρπούς των ειρηνευτικών αυτών σχεδίων και προγραμμάτων. Ξέρω περί τίνος πρόκειται. Έχω πολύ συγκεκριμένη αντίληψη θετική για την ενιαία πράξη η οποία άνοιξε τα σύνορα, τα οικονομικά ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες και περιοχές και η Ευρώπη πράγματι πέτυχε εδώ σε επίπεδο ειρήνευσης και συνεχίζει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη της ειρήνης στην Ιρλανδία γενικά ειρήνη, οικονομική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Γκάλαγκερ. Θέλει κανείς το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από χθε το βράδυ γνωρίζω πως είμαι η όντης για αυτό το θέμα από την πλευρά της μου πολιτικής ε, ομάδας, αλλά σε ό,τι αφορά αυτό το peace ε, program, το νευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο αυτής της περιφερειακής ε, πολιτικής ε, δεν ε, το κάνω για πρώτη φορά. Πάντοτε υποστήριζα αυτό το πρόγραμμα και τα όσα προτείνετε εσείς στην έκθεση αυτή, κύριε Κέλλη, τα υποστηρίζουμε και αυτά. Επειδή λοιπόν υποστηρίζουμε σε τέτοιο βαθμό αυτή την έκθεση δεν θα υπάρξουν και τροπολογίε από την πλευρά τη δική μα ε, πολιτική ομάδα. Θα πρέπει να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι πραγματικά υποστηρίζουμε εμφαντικά την ειρηνευτική διαδικασία στην Βορειοελλανδία και ότι ενδιαφερόμαστε για αυτή. Ε, στην ε, αιτιολογική, στο αιτιολογικό κομμάτι αναφέρεται κάποια παραδείγματα και ίσως θα μπορούσαμε να προτείνουμε και κάτι στην κατεύθυνση των βέλτιστων πρακτικών, των best practices. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε δηλαδή εδώ εσωτερικά μέσα στην ε, Επιτροπή μας ε, τι ακριβώς ήταν εκείνο που οδήγησε σε επιτυχία αυτό το πρόγραμμα. Γιατί ίσως και άλλες περιφέρειες ε, χρειάζονταν κάτι τέτοιο. Δεν επρόκειτο δηλαδή για ένα κανονικό αν θέλετε περιφερειακό πρόγραμμα. Επρόκειτο για ένα περιφερειακό πρόγραμμα με ιδιαίτερη σημασία και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Όχι. Τότε θα ήθελα και εγώ να πω κάτι, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια παρακολούθησε εκ του αυτή τη διαδικασία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της ειρήνης και της επανασυμφιλίωσης στην Βόρεια Ορλανδία. Και όπως είπε και ο κύριος Κάλεχερ, η ενίσχυση αυτή υπερβαίνει την ε, συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία. Γιατί έχουμε και το Ιντερεκ, το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας στο νησί της Ιρλανδίας, αλλά και το πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο συμμετέχει η Βόρεια Ιρλανδία. Επιπλέον όμως, <clears throat> μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το παρόν ε, και ως παρατηρήτρια στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία και είχαμε στενή συνεργασία με αυτό. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προηγούμενη, κοινοβουλευτική, στην προηγούμενη θητεία της ε, σύστησε μία διυπηρεσιακή ομάδα οριζόντια που κάλυπτε όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε στενή συνεργασία με την Ιρλανδία για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε όλα τα προγράμματα, ερευνητικά, ενεργειακά, προγράμματα μεταφορών, <clears throat> ώστε και οι αρχές και ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που είχαν για συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επιπλέον, όπως είπε και η Κωνσταντζα Κρέλ, σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της ε, Βόρεια Ιλλανδίας ε, ω υπόδειγμα καλής πρακτικής, αν όχι και για άλλα εδάφη. Και μάλιστα πριν από δύο χρόνια, στη διάρκεια των Open Days, είχαμε συνάντηση και με άλλες περιοχές, ε, με την Κύπρο, με τη χώρα των Βάσκων. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε το παράδειγμα της Βόρειας Ιλλανδίας για να προωθήσουμε και εκεί την συμφιλίωση γιατί υπάρχουν και άλλες ε, τέτοιες καταστάσεις ε, και το πρόβλημα υπερβαίνει το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία. Θα μπορούσαμε ίσως ε, να προσκαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμιά φορά συνεδρίαση για να μας παρουσιάσει την παρούσα κατάσταση και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στη Βόρεια Ιρλανδία. Είχαμε και ένα μαθητευόμενο από τη Βόρεια Ιρλανδία στο γραφείο μου και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και ο τωρινό Επίτροπος να διευκολύνει ε, την επικοινωνία μεταξύ της Ιρλανδίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Εδώ έχουμε μόνο δύο συναδέλφους από την Ιρλανδία, αλλά ανέκαθεν ναι, οι Ιρλανδοί ευρωβουλευτές ήταν πολύ δραστήριοι και υποστήριξαν ε, θερμά τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στην ε, Βόρεια Ιρλανδία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσει την πρόοδο που συντελέστηκε εκεί, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω δράσης. Και ευχαριστώ θερμά και το Σον και τους και γιατί χειρίστηκαν ε, και διεκπαιρέωσαν πολύ γρήγορα αυτή την έκθεση και είμαι βεβαία και στο μέλλον θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω για την έκθεση αυτή ότι άρχισε η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών που λήγει στις 5 Μαΐου το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση της, ομάδας, της Επιτροπής μας τον Ιούνιο και θα ξαναδώσω το λόγο στο Σον Κέλλη για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευγενική υποστήριξη που δείξατε προς το Ταμείο και στη διάρκεια της θητείας, της, της θητείας σας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάσουμε τα επιτεύγματα, γιατί πολλά έγιναν πραγματικά, όπως είπε και ο Πάτρε the Γκάλεχερ. Έχουμε πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα και τέτοιου είδους ειρηνευτικές διαδικασίες είναι πολύ εύθραυστες ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε, να θριαβολογούμε και να, να την κρίνουμε ως επιτυχή μια τέτοια διαδικασία. Μάλιστα πρόσφατα μια πολύ μικρή μειοψηφία το IRA έχει τοποθετήσει βόμβες σε διάφορα σημεία και μάλιστα τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός που έγινε θύμα, όχι επειδή ήταν στην αντίπαλη πλευρά, αλλά στην δική του, στο δικό του στρατόπεδο και να εκφοβήσουν άλλου από, τους, από το να καταταγούν στην αστυνομία. Γιατί στρατολογήθηκαν μέλη και από τις δύο πλευρές. Ήταν μια πολιτική 50-50% στελέχωση και αν προσπάθησαν να διαταράξουν αυτό το ποσοστό για να προκαλέσουν αναστάτωση. Γι' αυτό και είχαν στο στόχο στο κάποιον από το δικό του στρατόπεδο. Είναι έφρευστη η διαδικασία, θα, παραμείνει, θα παραμείνει έφρευστη ακόμη λίγο καιρό, όπω ήταν όλο τον τελευταίο χρόνο. Πάντω ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώ και είναι πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η εξέλιξη. Σα ευχαριστώ. Οπότε ολοκληρώνουμε το σημείο 7 τη ημερήσιας διάταξη και μια και μα περίσεψε λίγο χρόνο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα χθεσινά συμπεράσματα της συνεδρίας των συντονιστών. Οι συντονιστές έλαβαν τις εξής αποφάσεις. Καταρχήν, για τις ε, γνωμοδοτήσεις, οι συντονιστές αποφάσισαν να μην εκπονηθεί γνωμοδότηση επί της εκθέσεως ε, της ε, Επιτροπής Πολιτισμού για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Σήμα, το Ευρωπαϊκό Σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς, Αρμόδια κατ' ουσία, επαναλαμβάνει η, πολιτική, η Επιτροπή Πολιτισμού. Δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση για αυτό το θέμα. Δεύτερον, η γνωμοδότηση επί της προτάσεως κανονισμού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους κανόνες και γενικές αρχές των μηχανισμών ελέγχου των κρατών μελών για τις εκτελεστικές δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια κατ' ουσία νομική επιτροπή, αποφασίσαμε η γνωμοδότηση αυτή να εκπονηθεί από την Πρόεδρο και επίσης οι συντονιστές αποφάσισαν να μην εκπονηθεί γνωμοδότηση επί της εκθέσεως με θέμα τη σύναψη του πρωτοκόλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο στη σύμβαση για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις παράκτιες ε, περιοχές της Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας, έγινε μόνο η αρχή της συζήτησης και συμφωνήσαμε οι συντονιστές να αξιοποιήσουν τις επόμενες εβδομάδες και να διερευνήσουν τις διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν για να υποβάλουν προτάσεις μέχρι τα τέλη Μαΐου για θέματα ώστε αμέσως μετά να λάβουμε αποφάσεις για το ποιε εκθέσεις ίδια πρωτοβουλία θα εκπονήσουμε στο μέλλον. Η συζήτηση αυτή γίνεται επειδή τέσσερις εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλία και μία έκθεση περιφαρμογής ε, θα εκπνεύσουν τους επόμενους μήνες. Οπότε είναι ευκαιρία στις ομάδες σας να συζητήσετε αυτό το θέμα των εκθέσεων της πρωτοβουλίας μέχρι τα τέλη Μαΐου, ώστε τον Ιούνιο να λάβουμε αποφάσεις για το ποια θέματα θα μας απασχολήσουν. Μέσω του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεχτήκαμε μία πρόσκληση από την Βουλή των Βρυξελών την περιοχή Βρυξελών πρωτεβούσης με πρόταση της σύσταση ομάδας εργασίας μικτή με μέλη της ε, Βρυξελιώτικης Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της δικής μας Επιτροπής, προκειμένου να ετοιμαστεί η επόμενη συνάντηση. Αποφασίσαμε τελικά να μην δεχτούμε αυτό το αίτημα, γιατί είναι πάρα πολλές οι περιφέρειες της Ευρώπης και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιου είδους προσκλήσεις αν υποβληθούν από όλες τις περιφέρειες. Οπότε, ούτως ή άλλως, έχουμε τον Ιούλιο την ε, μεικτή συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και αυτό είναι το κατάλληλο φόρουμ για επαφές με τους Εθνικούς Βουλευτές. Γι' αυτό αποφασίσαμε να απορρίψουμε αυτή την πρόσκληση της Βουλής των Βρυξελών. Οι συντονιστές αποφάσισαν επίσης για τα πειραματικά προγράμματα στα πλαίσια του προπολογισμού του 2011. Αποφάσισαν οι συντονιστές να συστήσουν στα μέλη της Επιτροπής μας την υποβολή κάποιων θεμάτων για τα πειραματικά προγράμματα μέχρι τις 20 Μαΐου. Πρόκειται για μια προκαταρκτική διαδικασία που θα διευκολύνει τη διαχείριση των μελλοντικών πειραματικών προγραμμάτων. Πάντως, οι επίσημες αποφάσεις θα ληφθούν μετά το καλοκαίρι στα πλαίσια της κανονικής δημοσιονομικής διαδικασίας. Αυτή είναι μια προκαταρκτική διαδικασία που πρότεινε η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Καλό θα ήταν ε, και εμείς να εξετάσουμε αυτό το θέμα και να λάβουμε την απόφαση πριν τις 20 Μαΐου. Ο Λαμπέρτ Βανίστερ Ρόι έκανε μια πρόταση για τις Open Days και τη συνεργασία μας με την Επιτροπή των Περιφερειών. Η Γραμματεία θα ενημερώσει τους συντονιστές για τις πρωτοβουλίες και τις προετοιμασίες ό,τι αφορά τις Open Days και τις λεπτομέρειες ε, της συνεργασίας μας με την Επιτροπή Περιφερειών. Θα ενημερωθούν ε, το συντομότερο δυνατό οι συντονιστές και στη συνέχεια θα ενημερώσουν και τα υπόλοιπα μέλη. Αυτά δεν ήρθαν χθε στη συνεδρία των συντονιστών. Δεν ξέρω αν θέλει κανεί το λόγο. Μια και δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρώ ότι οι αποφάσεις των συντονιστών εγκρίθηκαν και από την Επιτροπή. Τώρα έχουμε ένα δίλημα. θα περάσουμε στη συζήτηση με την κυρία Βέστελ, γιατί μας έμεινε ένα τέταρτο μέχρι την έναρξη των ψηφοφοριών. Να ασχοληθούμε τώρα με το σημείο 13, την έκθεση κυρία Βέστφαλ, που κανονικά θα πρέπει να τη αφιερώσουμε μισή ώρα και να αρχίσουμε ένα τέταρτο αργότερα τι ψηφοφορίε. Ή να διακόψουμε μέχρι τι 10 για να αρχίσουμε τι ψηφοφορίε όπω προγραμματίστηκε στι 10. Καλύτερα να μην χάσουμε αυτό το τέταρτο Οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Βέστφαλ για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Ευχαριστώ. βέβαια θα είναι λίγο προβληματική η κατάσταση εάν δεν είναι εδώ η κυρία Σρότερ γιατί αναφέρεται στη δική της αγνομοδότηση και ε, η παρούσα αγνομοδότηση. Άρα προτείνω να αναβάλουμε λίγο αυτή τη συζήτηση γιατί σας λέω είναι και η συγκέντρια εκείνη τη γνωμοδότηση, ενδεχομένω να χρειαστεί να ξανακάνουμε τη συζήτηση. Αλλά βέβαια ίσω δεν την έχω δει εγώ την κυρία Σερότερα. Αν πρόεδρε δεν την βλέπετε ούτε εσεί, ε, θα ήθελα να βάλουμε λίγο τη συζήτηση. Ναι, βλέπω καλύτερα από εδώ, αλλά δεν βλέπω πουθενά την κυρία Σερότερα. Οπότε, εάν διαφωνεί κανεί, θα διακόψουμε προσωρινά. Αλλά ενδεχομένω θα μπορούσαμε να καλύψουμε τα τελευταία σημεία της σας διάταξης υπό τα διάφορα. Το ε, σημείο 15 της σας διάταξης υπάρχει κάτι. 15 ε, um, ε, λοιπόν το καλύψαμε. Ε, στις, στο σημείο 16 ημερομηνία της προσεχούς ε, συνεδρίασης σε 2 Ιουνίου λοιπόν, ε, 3 με 6.30 το απόγευμα και θα ήθελα να σας ζητήσω να μην αργήσετε. Σεβαστείτε εδώ τους χρόνους που έχουν προβλεφθεί, ούτως ώστε να προλάβουμε να κάνουμε αυτά που θα πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν μας έχει μείνει α, η ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σημείο 14 και η ψηφοφορία. Άρα λοιπόν διακόπτουμε τώρα μέχρι τις 10 και θα ξεκινήσουμε με τη ψηφοφορία εάν θα είναι δυνατό. Ελπίζω πως θα είναι δυνατό. Ακριβώς στις 10 να ξαναρχίσουμε. Διακόπτουμε λοιπόν για 15 λεπτά.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 Dear colleagues, can you check your machines now, so that we don't lose time later. Μπορείτε λίγο να ελέγξετε τα μηχανήματα της ψηφοφορίας που έχετε συνάδελφοι για να μην υπάρξουν προβλήματα αργότερα. Dear colleagues, we have technician, technicians with us now, so if anybody has problems... Έχουμε και τεχνικούς α, ε, για υποστήριξη και επειδή σήμερα θα χρειαστούμε τη, τα μηχανήματα, παρακαλώ ελέγξτε λειτουργούν μπροστά στις συσκευές. So, So can we, we open the votes? Can we check the votes? We open the votes. Λοιπόν, ελέγχουμε. Δοκιμαστή ψηφοφορία. η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Τρεις. Ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Μπορείτε, σας παρακαλώ όλοι να ψηφίσετε. εδώ αλλάζουν συνέχεια οι αριθμοί στην οθόνη. Τώρα νομίζω πως έχουν ψηφίσει όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. It works, I understand. So we can start voting. We start with point. Καλώς, ξεκινάμε λοιπόν με το ε, σημείο 8. Είχαμε ένα τροπολογίε οι οποίε είχαν κατατεθεί και κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε όπω προέκυψαν από τι διαπραγματεύσει. Ε, Ρικάρδο Κορτέ Λάστρα και στη διάσκεψη των Προέδρων ε, είχε υποστηριχθεί στις 14 Απριλίου η αλλαγή του τίτλου, οπότε σήμερα ε, ψηφίζουμε επί της έκθεσης σε ό,τι αφορά την ε, συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της στρατηγικής 2020 ε, στην ε, Ολομέλεια του Μαΐου θα έχουμε την ε, σχετική συζήτηση και την ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 10 και, 11. Ψήφι υπέρ. Αποσίες κατά. Εκκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποσίες. Ε, Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για τροπολογία 14 πάντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 λοιπόν ψήφι υπέρ, αλλά άρα εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές. Δυστυχώς δεν είμαστε σίγουροι, θα πρέπει να ψηφίσουμε ξανά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 15. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ και 16 κατά. Προφορική τροπολογία από τον εισηγητή για την παράγραφο 4. Θέλει να πάρει το λόγο εισηγητής. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 ψήφι υπέρ κατά και πάλι εδώ δεν είμαστε σίγουροι ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 18 ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας 22 ψήφοι υπέρ 14 κατά εγκρίνεται η 19 έχει αποσυρθεί 20 ψήφι υπέρ Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την τροπολογία 20. Άρχεται ψηφοφορία. 18 υπέρ, 19 κατά, άρα καταπίπτει. Τροπολογία 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 23 έχει αποσυρθεί 24 και 25 είναι ίδιες οπότε ψηφίζουμε και για τις δύο ψήφοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα συμβαστική τροπολογία 2 και την παράγραφο 11 που καλύπτει τις τροπολογίες 26 και 27. ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 για την παράγραφο 13 που καλύπτει τις τροπολογίες 29, 30, 32 και 34. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 όχι. Πάμε στην συμβαστική τροπολογία 4 για την 13α που καλύπτει τις 36 και 37 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 για την παράγραφο 13α που καλύπτει τις τροπολογίες 38 και 69 Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 39. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 40 έχει αποσυρθεί, οπότε περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 6. Παρακαλώ. σε ό,τι αφορά τη συμβαστική τροπολογία 6 θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση εδώ στην αγγλική μετάφραση Upland Regions λέμε εδώ εντάξει ορεινές περιοχές ε, στη γερμανική αλλά ίσως στα αγγλικά θα έπρεπε να αλλάξει η μετάφραση να λέμε Mountain Regions ορεινές περιοχές να ληφθεί αυτό υπόψη ε, στη μετάφραση ναι, ναι, συμφωνούμε μαζί σα σε όλα τα έγγραφα. Αυτή την έκφραση χρησιμοποιούμε. Mountain Regions. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη συμβαστική τροπολογία 6 που καλύπτει τι τροπολογίε 41 και 81. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαστε σίγουροι. Θα πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν για την τοπολογία 43. Ψήφι υπέρ άρχεται, ε, ψηφοφορία. The vote is closed. Πέραση της ψηφοφορίας. 24 ψήφι υπέρ, 18 κατά, άρα εγκρίνεται. Άρα καταβλήτη είναι 42. Πάμε σε 44. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για τη 44 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας 16 υπέρ 24 κατά άρα απορρίπτεται. Η 45 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 47 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται. Η 46 καταπίπτει. Πάμε στη 48 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεν γνωρίζουμε, άρα λοιπόν θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 48. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 18 ψήφοι υπέρ και 24 κατά. Συμβαστική τροπολογία 7 στην παράγραφο 15α που καλύπτει τις ε, τροπολογίες 49 και 51. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 8 που καλύπτει την, τις ε, τροπολογίες 52, 53 και 54. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τροπολογία 50 που έχει αποσυρθεί. Κατά. Ε, πάμε λοιπόν στη 55. Αν καταπίπτει αυτή, οπότε πάμε στη τροπολογία 57, καθώς και 56 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 57 λοιπόν, ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. Για την 57 λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της 23 υπέρ 18 κατά, άρα εγκρίνεται τελικά. Τροπολογία 58, ψήφι υπέρ. Κατά. Πολύ δύσκολα και εδώ να εμπιστώσουμε το αποτέλεσμα, άρα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Μεταξύ της ψηφοφορίας, πέρας της 18 υπέρ 23 κατά. Άρα λοιπόν Απορρίπτεται. Πάμε στην 59. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Είναι σαφέ. 60. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 61. Πέραση ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 18 ψήφι κατά, άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 62, ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται, 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 64 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 67 και 68 66 λοιπόν υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε για την 66 λοιπόν Πέραση τη ψηφοφορίας, 24 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 67 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είμαστε σίγουροι, ψηφίζουμε για την τροπολογία 68. Πέραση τη ψηφοφορίας, 18 ψήφοι υπέρ, 23 κατά, άρα απορρίπτεται. 69 καταβίπτει. 70 ψήφοι υπέρ, κατά. Αποχές. Είναι σαφές ότι απορρίπτεται, έτσι δεν είναι. 71 ψήφοι υπέρ, κατά. Αποχές Απορρίπτεται 72. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε για την τροπολογία 74. Πέρας της ψηφοφορίας 25 ψήφοι κατά, 16 υπέρ, άρα απορρίπτεται. 75 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 για την παράγραφο 21 που καλύπτει τις τροπολογίες 78 και 79 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε μετά στη συμβαστική τροπολογία 10 που καλύπτει τις ε, τροπολογίες 80, 82 και 83. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 84, τροπολογία 84. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε για την τροπολογία 85 έναρξη της ψηφοφορίας, πέρας της ψηφοφορίας, 28 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 86, ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 για τις τροπολογίες 89, 90 και 91 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την τροπολογία 92, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έναξη λοιπόν της ψηφοφορίας, πέραση της ψηφοφορίας, 24 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 93, ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94. Πνευματική ψηφοφορία που ζητήθηκε από την συγκίτρια για το πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα, δεύτερο κομμάτι της τροπολογίας 94, έναρξη της ψηφοφορίας. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται 23 ψήφι υπέρ ενάντια 14 ψήφων κατά και 4 αποχών. 95 έχει αποσυρθεί. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 26 έχουμε μια προφορική τροπολογία από την κυρία που ε, δεν είναι εδώ αλλά μπορεί να την εκπροσωπήσει κάποιος. Ψηφίζουμε λοιπόν για την προφορική τροπολογία για την παράγραφο 26. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 98. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε. Νομίζω. Για την 97. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ και 17 κατά. Τροπολογία 99 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στα εκτιμώντας. Τροπολογία 1 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε σε βασική τροπολογία 1 για το εκτιμώντα D που καλύπτει τι τροπολογίε 7 και 8. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 9. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ θα ελέγξουμε για την τροπολογία 9 σε σχέση με το εκτιμώντας Dα. Α. της ψηφοφορία, πέραση της 25 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, άρα εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία για το σύνολο δηλαδή θα γίνει ηλεκτρονικά για το σύνολο του σχεδίου έκθεσης. Πέραστης τη ψηφοφορία. 40 ψήφοι μία ψήφος κατά και μία αποχή. Άρα λοιπόν, ε, υιοθετείτε παρούσα έκθεση, συγχαρητήρια. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Just one question. Μία ερώτηση. Όταν ξεκινήσαμε την ψηφοφορία, είπατε ότι θα μπει στην ημερήσια διάταξη του Μαΐου. Θέλουμε κατά προτεραιότητα συζήτηση μερικών εκθέσεων πρωτοβουλία. Αλλιώ απλώ ακούμε μια παρουσίαση του εισηγητή μόνο ή το Μάιο ή τον Ιούνιο, αλλά να έχουμε κατά προτεραιότητα συζήτηση για τη συνοχή. Γιατί έχουμε και άλλες εκθέσεις, γιατί να μην τις προωθήσουμε με συζήτηση. Δεν ε, έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις. Κατά πάσα πιθανότητα η έκθεση του Ρικάρντο Λάστρα ίσως περάσει στην Ολομέλεια του Μαΐου. Και φυσικά το έχουμε ζητήσει για όλες μας εκθέσεις, όχι μόνο για μία, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη το αποτέλεσμα, δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις. Επίσης δεν είναι σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ε, συνεδρίασης του Μαΐου. Μπορεί η συζήτηση να γίνει στην πρώτη και η, η ψηφοφορία στη δεύτερη. Πάντως νομίζω ότι η συζήτηση θα γίνει στην πρώτη συνεδρίαση του Μαΐου. Um, Κωνσταντζα Κρέλ. Ναι, και στο ΕΛΚ αυτό συζητήσαμε και στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών και θα προτείνουμε συζήτηση κατά προτεραιότητα της πολιτικής συνοχής στη δεύτερη ολομέλεια του Μαΐου. Αυτό είχαμε ζητήσει. As we decided we have... Αυτό είχαμε αποφασίσει και αυτό είχαμε ζητήσει να εξεταστούν και οι δύο εκθέσεις μας στην Ολομέλεια με συζήτηση κατά προτεραιότητα. Συνοχή και στρατηγική του 2020. Είναι αναφυσβήτητο ότι θα περάσει με συζήτηση κατά προτεραιότητα η έκθεση του Ρικάρντο Κορτέ Λάστρα, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση επίσημα. Πάντως το ζητήσαμε και στη συνδιάσκεψη των Προέδρων. Και για τη δική σας έκθεση είμαι σχεδόν σίγουρη, αλλά για τις άλλες κρεμούν οι αποφάσεις. Πάντως δίνουμε μάχη για να περάσουν όλες με συζήτηση κατά προτεραιότητα. Και θα ήθελα είτε επίσημα είτε ανεπίσημα να ασκήσουμε πίεση και στις πολιτικές ομάδες γι' αυτό. Γιατί γιατί τελική απόφαση τη λαμβάνει η διάσκεψη των Προέδρων. Οπότε έχει σημασία η πολιτική υποστήριξη, υποστήριξη από τις πολιτικές ομάδες. Ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα. Για να περάσουμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Την έκθεση του Λάμπερτ Βαν Ρόι για την υλοποίηση των συνεργειών των πόρων που προορίζονται για την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες. Κατατέθηκαν 74 τροπολογίες, πολλές δηλαδή, και μάλιστα η έκθεση εκπονήθηκε με βάση το, το άρθρο 50 σε συνεργασία με άλλες επιτροπές Έχετε λάβει το κατάλογο ψηφοφορίας και μπορούμε να αρχίσουμε. Συμβαστική τροπολογία 1 που καλύπτει τις τροπολογίες 6, 7 και 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Η 9 έχει αποσύρθει. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 που καλύπτει τις τροπολογίες 12, 16 και 53. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Ή όχι. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Τροπολογία 50 παρακαλώ συνάδελφοι. Και θα ψηφίσουμε κατά τμήματα, όπω ζήτησε το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική Προφορική τροπολογία τώρα. Ποιος είναι υπέρ. It is ε, carried. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 με την προφορική προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. 21. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 που καλύπτει τις τροπολογίες 17, πρώτο τμήμα της ΙΤΡΕ παράγραφος 4, 24-26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 έχει αποσυρθεί 27 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 15 πρώτο τμήμα είναι κατά τμήματα η ψηφοφορία ψηφίζουμε το πρώτο ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Προφορική τροπολογία του εισηγητού για την 29. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Την 29 όπως έχει τροποποιηθεί από την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8, πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 που καλύπτει τις τροπολογίες 30, 31, 46 και την παράγραφο 12 της ΙΤΡΕ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 που καλύπτει την παράγραφο 9 της ΙΤΡΕ, δεύτερο τμήμα της παράγραφου 15 ΙΤΡΕ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 35 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Πρώτο τμήμα. Α, συγγνώμη, έχει εγκριθεί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 Απορρίπτεται 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 που τις τροπολογίες 11, 44, 45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 αποκαλύπτει τις τροπολογίες 48 και δεύτερο τμήμα της 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία στη 49 από την κυρία Κρέλ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 που καλύπτει τις τροπολογίες 51, 52, 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 54. Άρχεται η ψηφοφορία. The Ψηφίζουμε την 54. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψήφισαν 15 υπέρ και 24 κατά, άρα απορρίπτεται. 55. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. Η 56 καταπίπτει. 57 ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. Τέλος. 13 ψήφισαν υπέρ και 27 κατά, άρα απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 αποκαλύπτει τις τροπολογίες 63, το δεύτερο τμήμα της Ήτρε παράγραφος 4. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 64. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 66 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική τροπολογία 14 που καλύπτει τις τροπολογίες 67, 68, 69, την παράγραφο 5 της Ήτρε, πρώτο τμήμα της 6 Ήτρε. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14 έχει εγκριθεί χωρίς ψηφοφορία. Τροπολογία 70. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15 για δεύτερο τμήμα της παραγράφου 6 της Ήτρε, δεύτερο τμήμα της 11. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 προφορική τροπολογία του συγητού. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 τώρα πώς έχει τροποποιηθεί. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 έχει εγκριθεί χωρίς ψηφοφορία. 74. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Πρώτη αποσύρεται, δεύτερη τροπολογία, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τρία έχει αποσύρθει, τροπολογία τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1, καταπίπτει. Τροπολογία 5, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία της έκθεσης του Λάμπερτ Βανίστερ με ηλεκτρονικό τρόπο παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ. Μία ψήφος κατά και μία αποχή. Colleagues, you need a break Μήπως θέλετε διάλειμμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Όχι. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία της έκθεσης για τη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και τη χρηματοδότησή της. Ο κύριος Στρεμόπουλος θέλει να πει κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Εξακολουθείτε να θέλετε το λόγο. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Έχουμε 54 ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει τον Ιούνιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία υπαριθμών 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ε, Περνάμε στην 7. Στην προφορική στην 7. Υπέρ. Κατά. Εσ. Δεκτή. Τώρα κανονικά την 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8. Έχουμε την προφορική πάλι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ποιοι είναι. Θα πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Για μια στιγμή. Περιμένετε. Μια στιγμή. Ψηφίσαμε υπέρ της τροπολογημένης 8. Περνάμε τώρα στην 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την ενέα ζητώ συγγνώμη αλλά πρέπει να ελέγξουμε. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 11. 28 υπέρ, 13 κατά. 12 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13. 13 και 14 ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Περνάμε στη συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εικοσιτέσσερα. με προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 25 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 26 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 27 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 28 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές απορρι... Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 30. Τέλος. 27 υπέρ 13 κατά. Υπάρχει μια διάσπαση ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες και είναι δύσκολο να μπορέσω να κρίνω εύκολα από την ανάταση των χείρων. Λοιπόν, 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές αν νομίζω ότι απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σαφές. Η 37 καταπίπτει.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 Τέλος της ψηφοφορίας. 27 υπέρ 11 κατά. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες πλέον για το αποτέλεσμα. Πηγαίνουμε τώρα στην 36. Σταματήστε να σχολιάζετε, λέει η πρόεδρος. 36. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, σαφές. 39. Ψήφος κατά διέρεση. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 40 έχει αποσυρθεί. 41 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή, αλλά μήπως θέλετε να ελέγξουμε. Όχι, γίνεται δεκτή, δεν υπάρχει αμφιβολία. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Δεν σηκώνετε πλέον τα χέρια σας. Πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν για την 43. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται 17 υπέρ 22 κατά. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 50 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 51 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 52 έχει αποσυρθεί. 53 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι γίνεται δεκτή. Ελέγχουμε την 53 ηλεκτρονικά. 53. Λοιπόν, 27 υπέρ 11 κατά. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τρίτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέταρτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην τελική ψήφο. Άρχεται η ψηφοφορία, η ηλεκτρονική ψήφος. «34 υπέρ, 1 κατά δύο αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Uh, Ανακοίνωση της ε, Επιτροπής για την πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Έχουμε και τέσσερις συμβιβαστικές τροπολογίες. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα γίνει στις 30 Μαΐου ή 31 Μαΐου δεν άκουσα. Λοιπόν, τροπολογία 3, ξεκινάμε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ένα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Πέντε υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε στην 8 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 1. Αποκαλύπτει την... Α, θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Θα πρέπει να ελέγξουμε για μια ακόμη φορά γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα. Όλοι είναι υπέρ λοιπόν, όλοι όμως. Λοιπόν, συμβιβαστική υπαριθμένα. Υπέρ, κατά, δεκτή. Δύο, υπέρ, κατά, δεκτή σαφώς. Στην 14 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 18 υπέρ, κατά, αποχές, Δεκτή. Περνάμε τώρα στην τρίτη συμβιβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 22 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στη συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή έχουμε τώρα την προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4 δέλτα μικρό του πίπα ψηφίζουμε και είναι υπέρ κατά, αποχές, δεκτή η προφορική τροπολογία Πίπερ. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και 30 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα το, το ψήφισμα. ηλεκτρονική ψηφοφορία. ...37 υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες λοιπόν. Συγχαρητήρια. Δεν έχουμε διάλειμμα συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Δεν έχουμε διάλειμμα, επαναλαμβάνω. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Βέστφαλ. Όσοι θέλετε να κάνετε συζητήσεις εκτός εθούσης παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, αγαπητοί κύριε και κύριοι συνάδελφοι, να σας εξηγήσω γιατί δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε προηγουμένω ε, την ε, γνωμοδότηση όταν δεν ε, βρισκόταν εδώ η κυρία Σούχετα. Η δική μας λοιπόν νομοδότηση ασχολείται και αφορά πάρα πολύ τη δική της νομοδότηση από την Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων, οπότε α, προφανώς έπρεπε να βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, η Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων ασχολείται με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, δηλαδή το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία την, το δυναμικό της απασχόλησης. Ε, μας κάνει λοιπόν κάποιες προτάσεις σε ό,τι αφορά φιλοπεριβαλλοντικές ε, θέσεις εργασίας, θέτει ερωτήματα σε ό,τι αφορά το δυναμικό της απασχόλησης και θέτει ερωτήματα σε σχέση με την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να εργάζονται σε φιλοπεριβαλλοντικές, σε πράσινες θέσεις εργασίας οι πολίτες. Ε, θεωρούμε πως μια τέτοια γνωμοδότηση είναι χρήσιμη καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η πράσινη οικονομία λαμβάνει μεγαλύτερη σημασία και αυτό βρίσκει σύμφωνος ε, και τους σοσιαλδημοκράτες. Ε, Εμεί, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δική μα νομοδότηση τη ε, Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, δεν επισέρχομαι σε επιμέρου με αυτή τη νομοδότηση. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να προσπαθήσω να σκεφτώ ποιες ιδέες μπορώ εγώ να εισάγω σε αυτή τη γνωμοδότηση από την πλευρά της ε, Επιτροπής ε, ε, Περιφερειακής Πολιτικής, αλλά επειδή είχα μόνο 1500 χαρακτήρες στη διάθεσή μου, τόσο ώστε να αναπτύξω τη δική μας θέση, περιορίστηκα σε κάποια σημεία προτεραιότητας. Καταρχήν, τα διαφορετικά ταμεία παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Οι περιφέρειες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας μπορούν πράγματι να ε, βασιστούν στην υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωση, ειδικότερα στον χώρο της ε, παιδείας, η οποία όπως γνωρίζουμε αποτελεί τη βάση για την απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων, οι περιφέρειες και οι δήμοι και κοινότητε έχουν ε, πολλά κοινά. Οι γενικότερε συνθήκε για την περαιτέρω κατάρτιση βρίσκονται στον χώρο τη ευθύνη των διάφορων περιφερειακών φορέων και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ε, στις οποίες συγκαταλέγεται ή ε, για παράδειγμα ε, επέκταση της, των διάφορων τοπικών συγκοινωνιών και μέσω μεταφοράς. Η αυτό το στοιχείο, όπως αναφέρεται και στην γνωμοδότηση της κυρία Σρότερ, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ε, για όλους ε, ψάχνουν εργασία. Η κινητικότητα δηλαδή ε, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του ώστε μπορεί κανείς να μεταβεί στο σημείο που λαμβάνει την εκπαίδευση στη θέση εργασίας. Και οι τοπικές ε, ε, συγκοινωνίες είναι πολύ σημαντικές εδώ γιατί ε, οι πολίτες εκείνοι οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους έχουν ένα κατάλληλο δίκτυο τοπικών συγκοινωνιών μπορούν να μεταβούν εύκολα στις θέσεις εργασίας τους και κατά συνέπεια τόσο εδώ όσο και στον στο χώρο της εκπαίδευσης είναι, απαραίτητο είναι απαραίτητος ο εξυγχρονισμός των αντίστοιχων υποδομών ώστε να υπάρξει και μια ταυτόχρονα υποστήριξε από, την, από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο θίγω στη δική μου γνωμοδότηση είναι η βιωσιμότητα των διαρθρωτικών ε, πόρων. Εγνωρίζουμε δηλαδή όλη τις περιπτώσεις εκείνες όπου ε, διάφορες επιχειρήσεις έχουν ε, λάβει χρηματοδοτήσεις από τη διαρθρωτικά ταμεία για να δημιουργήσουν νέες μονάδες παραγωγής τις οποίες όμως μετά εγκαθιστούν αλλού μετά από ορισμένα χρόνια. Πράγμα το οποίο είναι προβληματικό γιατί εμείς θέλουμε να δημιουργούμε βιώσιμες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ε, λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας την βιωσιμότητα, δηλαδή τον πρόθεσμο χαρακτήρα συγχρηματοδοτούμενων έργων. Αυτά τα κονδύλια δηλαδή θα πρέπει να παραμένουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να επενδύουμε σε επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν μόνο για μικρό χρονικό διάστημα κάποιες θέσεις εργασίας και μετά μετεγκαθιστούν αυτές τις θέσεις εργασίας αλλού. Επίσης, αναβαίνω ε, στη γνωμοδότησή μου και το πρόγραμμα Εράσμους για τους ε, τοπικούς και περιφερειακούς αντιπροσώπους. Ε, ακόμα και αν σε αυτή τη φάση δεν είναι σαφές το ποια συνέχεια θα δοθεί σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά παρόλα αυτά αυτό το πρόγραμμα είναι σίγουρο πως μπορεί να δώσει περαιτέρω ευκαιρίες και να βοηθήσει τις περιφέρειες στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών τους. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, την πολιτική για την αγορά εργασίας μπορούν πολλά να μάθουν από αυτό το πρόγραμμα οι ε, πρόσωποι μας στο περιφερειακό επίπεδο. Και Άκουσα από τον κύριο Χάν ότι βρίσκεται στο πλευρό μας σε ό,τι αφορά δηλαδή την περαιτέρω ανάπτυξη του πρόγραμματος Εράσμους. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για την πρώτη ονομοδότηση την οποία έχω συντάξει εγώ και ελπίζω να έχω πράγματι συμπεριλάβει εδώ τα κυριότερα σημεία από την πλευρά δηλαδή της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Πολιτικής και να βοηθήσω την κυρία Σόντερ στη δική της γνωμοδότηση. Αναμένω λοιπόν ε, τώρα ε, τα σχόλια των συνδέων των και των συναδέλφων και θα ήθελα να ακούσω τι έχουν να πούν. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρο. Ε, να δώσουμε λοιπόν το λόγο τώρα στου υπόλοιπου στιώδη ε, Σκιώδη εισηγητέ. Ε, κυρία Σότερ είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την εισηγητρία για την πρώτη παρουσίαση ε, της ε, γνωμοδότησής της ε, και για την, το έργο που έχει καταβάλει εδώ. Εμείς βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό σε επαφές και έχουμε συζητήσει αυτή τη γνωμοδότηση. Μιλάμε για μια γνωμοδότηση πρωτοβουλία από την πλευρά της Επιτροπής Απασχόλησης, η οποία όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιατί προφανώς εδώ τίθεται διάφορε παράμετροι, αν θέλετε, από τη δική μα επιτροπή ω προ το πώ μπορεί να αξιοποιηθεί ένα τέτοιο δυναμικό στην απασχόληση. Τώρα, πώ διαρθρώνεται η γνωμοδότηση και πώ μπορεί να συμβάλλει η γνωμοδότηση αυτή εδώ τη επιτροπή ε, ε, σε εκείνη τη γνωμοδότηση. Η δική μα ε, γνωμοδότηση σχετίζεται με την πρωτοβουλία ότι η στρατηγική 2020 μας λέει ότι ναι θέλουμε να έχουμε αυτή την οικολογική αν θέλετε καμπή Πράγμα όμως τον οποίο δεν απηχείται καθόλου ε, στον τομέα της ε, απασχόλησης. Οι προεδρίες όμως, ε, όπως για παράδειγμα η Ισπανική Προεδρία με το New Skills for News Jobs, αλλά και άλλες προεδρίες έχουν θέσει εδώ την προτεραιότητα. Η Βελγική Προεδρία θα ήθελε να θέσει στο επίκεντρο τα green jobs, δηλαδή τις πράσινες θέσεις εργασίας και βρισκόμαστε σε επαφές με τις αντιστοιχές προεδρίες στην Επιτροπή. Απασχόλησης ε, και Κοινωνικών Υποθέσεων ε, εξέτασα 20 διαφορετικές ε, μελέτες σε διεθνές επίπεδο και είδα πως και σε σχέση με το G20 και στο G8 συζητείται επισταμένως αυτό το ζήτημα και για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον ορισμό των πρασίνων θέσεων εργασίας, των green jobs έχουμε λάβει εδώ την, ε, το σχετικό ορισμό που είχε ε, προταθεί και στους Υπουργούς ε, του G8. Και από αυτές τις μελέτες που εξέτασα διαγράφεται κάτι με σαφήνεια, ότι δηλαδή οι διάφορες γενικέ ε, συνθήκε, αν θέλετε, γενικέ προποθέσει είναι εκείνε που καθορίζουν το κατά πόσο αξιοποιείται το σχετικό δυναμικό. Υπάρχουν δηλαδή οι κατάλληλε συνθήκε, ούτω ώστε να μεταβούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ε, οι επενδυτέ και να πούνε ναι, αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε εδώ. Υπάρχει ένα σταθερό πολιτικό πλαίσιο. Ε, και σε ό,τι αφορά αυτό το σταθερό πολιτικό πλαίσιο, έχουμε διαπιστώσει πράγματι ότι στα, στα σημεία εκείνες περιοχές εκείνες όπου ασκείται σταθερή ε, πολιτική έχουμε επιχειρήσει να μεταβαίνουν εκεί κατά εκατοντάδες ενώ υπάρχουν άλλες ε, ε, περιοχές όπου αυτό δεν συμβαίνει για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή, την ενεργειακή, την απόδοση των διαφόρων εγκαταστάσεων και ούτω καθεξής. Όταν δηλαδή υπάρχει, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν σαφείς και σταθερές ε, παράμετροι σε ό,τι αφορά το γενικότερο πλαίσιο, δεν μεταβαίνουν εκεί οι επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια γενική πολιτική, μια δημοσιονομική πολιτική, ένα mainstreaming, μια δηλαδή ευθυγράμμιση των γενικότερων ε, πολιτικών ε, που θα λέει για παράδειγμα ότι επιθυμούμε την περαιτέρω ανάπτυξη των τομέα των επιχειρήσεών μας, της βιομηχανίας μας, της πόλης μας, της περιφερειάς μας. Και όπως αναφέρθηκε ήδη, η πόλη αποτελεί αν θέλετε ένα πυρήνα, μια συγκέντρωση ευκαιριών. Είτε πρόκειται για καλύτερη ενεργειακή απόδοση ε, κτηρίων, είτε ε, για κινητικότητα, είτε κινητικότητα που σχετίζεται σε σχέση με το κλίμα. Εάν μια πόλη πει ότι εμεί θα ασχοληθούμε με αυτό, αυτόματα προετοιμάζεται και η υποδομή. Για παράδειγμα, ε, δρόμοι, λωρίδες ε, για τα ποδήλατα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εφόσον δημιουργείται μια τέτοια υποδομή, προσέρχονται, προσελκύονται και αντίστοιχε επιχειρήσει και έτσι δημιουργείται ένα πυρήνα καινοτομία, ένα κλάστερ ε, καινοτομία υπάρχουν εδώ διάφορες εκτιμήσεις, ε, διάφορες τιμές ότι δηλαδή ε, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις που είναι θετικές και λένε ότι πράγματι όταν υπάρχουν κάποιε ορισμένε γενικέ προποθέσει, υπάρχει επιτυχία, ενώ υπάρχουν και αρνητικέ εκτιμήσει. Δηλαδή όταν δεν υπάρχουν τέτοιε προποθέσει, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ε, και την έκθεση του κ. Βανίστα πολύ σημαντική ως προς το σημείο δηλαδή του πώς μπορούμε να συσχετίσουμε αν θέλετε την έρευνα με την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εάν θέλουμε, για παράδειγμα, όταν λέμε ότι θέλουμε η οικολογική ανάπτυξη να αντιδράσουμε κάποιο τρόπο στις ε, κλιματικές μεταβολές, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα μπορέσουμε αυτό να το, ε, ε, να το αξιοποιήσουμε μέσα στις περιφέρειες, τι μπορούμε δηλαδή εδώ να κάνουμε σε επίπεδο καινοτομία. Κάτι τέτοιο έχει άμεσο αντίκτυπο ε, και στην αξιοποίηση του δυναμικού σε ό,τι αφορά την απασχόληση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και γι' αυτό θεωρώ πως αυτή η έκθεση είναι πολύ θετική, γιατί απηχεί ακριβώς αυτή τη διάσταση. Για μένα λοιπόν είναι σημαντικό η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να τροφοδοτήσει αυτή τη διάσταση, δηλαδή την περιφερειακή ε, διάσταση, ούτως ώστε στην Επιτροπή Απασχόλησης να διασφαλίσει ότι ε, θα αποτελέσει αυτή η διάσταση ένα χωριστό κεφάλαιο. Και να μην χρειάζεται ε, να κάνουμε και διαπραγματεύσει να ψηφίσουμε σχέση με αυτό το σύνολο ξεχωριστά. Να πούμε ότι ναι, αποτελεί μια ξεχωριστή διάσταση. Και θα το συζητήσουμε και περαιτέρω με την κυρία Βέσφα, αλλά έχουμε ήδη συζητήσει και προηγουμένως ελπίζουμε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να συμφωνήσουμε με αυτή την προσέγγιση και εκείνο που έχει εδώ ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ε, θα πρέπει ένα κομμάτι των διαρθρωτικών ταμείων να ε, επενδυθεί ακριβώς σε αυτή την οικολογική αν θέλετε μετάβαση, σε αυτή την πράσινη μετάβαση γιατί ε, τέτοιου είδου ε, οικολογικές ε, πρωτοβουλίε δημιουργούν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Αυτό έχει αποδειχθεί. Και σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει δεν έχουμε αντίστοιχη αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν έχουμε δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει άλλο κάνει το λόγο, άλλοι εισηγητές ή σκιώδη εισηγητές, γιατί δεν δηλώσετε ενδιαφέρον. Ο κύριος Βλάσακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που η συγκεκριά μας αναφέρθηκε στις αστικές μεταφορές και στο δυναμικό δημιουργία θέσεων απασχόλησης που εμπεριέχουν, γιατί πιστεύω ότι εκεί υπάρχει τεράστιο χρησιμοποιητό δυναμικό. Και αυτό είναι προτεραιότητα για τους περισσότερους δήμους και τα αστικά κέντρα. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό σχεδίων αλλά δυστυχώς πενιχρά κονδύλια στη διάθεσή μας. Γι' αυτό και καλό θα ήταν να ζητήσουμε από τους Δήμους και τις κυβερνήσεις να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια. Γιατί αν θέλουμε να υποστηρίξουμε κάποια προγράμματα και σχέδια, χρειαζόμαστε και τα απαραίτητα κονδύλια. Για την αγορά νέων οχημάτων, για παράδειγμα, και όχι μόνο για την κατασκευή υποδομών. Και θα πρέπει να ελέγξουμε τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδύλιων φυσικά. Το πρόγραμμα Έρασμος για τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους είχε παρκή κονδύλια. Παρ' όλα αυτά δεν απορροφήθηκαν πλήρως. Και μέχρι στιγμής ε, μόνο μια μελέτη εκπονήθηκε. Δεν καταφέραμε δηλαδή ακόμη να στείλουμε τοπικούς ε, αντιπροσώπους ή περιφερειακούς αντιπροσώπους σε πρόγραμμα ανταλλαγών το μας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ ο κύριος Λαμπέρτ Βαν Νίστελ Ρόι. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά και την εισηγήτρια για το έργο της. θα πρέπει να συνδέσουμε αυτή την έκθεση με την ε, εδαφική διάσταση των πρωτοβουλειών στα πλαίσια της φιλοπεριβαλλοντικής πράσινης οικονομίας. Κατά τη γνώμη μου, η στρατηγική του 2020 έχει πιο φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση. Αν όμως δεν υπάρξει και περιφερειακό όραμα ή περιφερειακή δημοτική διάσταση, Νομίζω ότι θα στοχίσουμε. Χρειαζόμαστε μια περιφερειακή διάσταση. Θα πρέπει να δώσουμε ναύσματα στην απασχόληση χάρη σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένα περιεκτικό όραμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να περιλάβουμε και την εδαφική διάσταση και την ανάγκη της ολοκληρωμένης προσέγγισης ε, στη χρήση των κονδυλίων μας. Δεύτερον, ανάγκη συντονισμού των διαφόρων επιπέδων και εναρμόνιση. Έτσι θα βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα αν έχουμε καλύτερη εναρμόνιση των δημοτικών πρωτοβουλειών με τις περιφερειακές και τις εθνικές ή και υπερεθνικές. Χρειάζεται λοιπόν ένας καλύτερος συντονισμός. Το βλέπουμε αυτό και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ηλεκτρικά οχήματα. Και εδώ βλέπουμε ότι κάθε πόλη επεξεργάζεται το δικό της σχέδιο, αλλά δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των πόλεων. Σίγουρα είναι απαραίτητες πιο αποκεντρωμένες πρωτοβουλίες αλλά και μια καλύτερη εστίαση και πιο έντονο συντονισμός. Εσείς ε, είχατε περιορισμό τους 1500 χαρακτήρες, ίσως θα μπορούσαμε με τις τροπολογίες μας να εμπλουτίσουμε την έκθεση, αλλά ήδη εσείς ε, θεσπίσατε τις πιο σημαντικές προτεραιότητες. Εμείς απλώς θα τις διανθίσουμε. Συγγνώμη, ο κύριος Κόβατσεκ, ε, ο συντονιστής του ΕΛΚ, δεν σας είδα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια για τις προτάσεις και το σχέδιο γνωμοδότησης. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους ότι και οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα αυτά και μάλιστα όταν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα καταρτίζουν σημαντικά έγγραφα στρατηγικής όπως αυτό για το 2020 και την κινητικότητα δεν θα πρέπει να παραμελούν την κινητικότητα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την πράσινη οικονομία. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ παλιών και νέων χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος οι νέες χώρες ό,τι αφορά και τις υποδομές και τις υλικές και τις τεχνικές. Αναφέρθηκε ο στόχος της ε, κοινωνίας με πλήρη απασχόληση. Εγώ έζησα τα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος και του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπου εκεί η πλήρης απασχόληση ήταν πραγματικότητα, αλλά κάπως αφηρημένη. Διαρωτώ με λοιπόν αν όντω είναι εφικτή μια κοινωνία πλήρους απασχόλησης. Μήπως καλύτερα να βρούμε μια πιο δόκιμη διατύπωση. Ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε, ε, κυρία Πρόεδρε ε, ορισμένες παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν, ε, ε μου κάνει κάπως εντύπωση η τοποθέτηση της κυρίας Βεστάλ για το θέμα που συζητάμε από την εξής άποψη. Εάν μέχρι στιγμή δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα της μαζικής μεταφοράς ε, των νέων και των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς, δεν ξέρω τι θα το κάνουμε τώρα με την πράσινη οικονομία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ε, ας είναι. Υπάρχει πρόβλημα ε, όντως και ειδικότερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπως ε, οι νέες χώρες όπως λέμε. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα σοβαρό, αλλά δεν έχει τόσο σχέση νομίζω εγώ με το θέμα που συζητάμε. Τι όμως νομίζω ότι ε, είναι ανάγκη να πάρουμε υπόψη μας. Καταρχήν κυρία Πρόεδρε δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι πολύ μεγάλα κεφάλαια θα στραφούν στις ε, πράσινες οικονομίες γιατί ελπίζουν από εκεί να βγουν από την κρίση του καπιταλιστικού συστήματος ε, που περνάει αυτή τη στιγμή. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι τόσο ε, να πούμε και εμείς κάτι για την πράσινη οικονομία, αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως. Εξάλλου δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, ε, την προηγούμενη εβδομάδα η Frankfurt Allgemeine Zeitung δημοσίευε ένα στοιχείο που δείχνει πόσο έχει προχωρήσει η Κίνα παραδείγματος χάρη στις τεχνολογίες αυτές της εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τη Γερμανία, στις παγκόσμιες αγορές και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα της Κομισιόν. Τα υπόλοιπα τώρα είναι κάπως δευτερεύοντα. Ε, θέλω να πω δηλαδή κυρία Πρόεδρε ότι αν ε, αυτή η στρατηγική θα εξακολουθεί να βασίζεται στο κέρδος και προφανώς αυτό θα εξακολουθεί να βασίζεται τότε τα όσα θέλουμε ε, να υλοποιηθούν όσον αφορά την απασχόληση και άλλοι τέτοιοι κοινωνικοί στόχοι δεν θα είναι δυνατοί. Αλλά για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Σωστό είναι αυτό που υπόθηκε ότι εν πάση περιπτώσει οι πόλεις αποτελούν πράγματι ένα τομέα και ε, αξιοποίησης των πράσινων ε, τεχνολογιών αλλά και ε, επιχειρήσεων για να δραστηριοποιηθούν. Όμως δεν είναι μόνο οι πόλεις. Παραδείγματο χάρη, νομίζω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να δούμε πώ θα το αντιμετωπίσουμε είναι το γεγονό ότι στην περιφέρεια, και εννοώ τώρα στην Ελλάδα εν προκειμένου αλλά και σε άλλε χώρε, θα εγκατασταθούν πολύ μεγάλε μονάδε ε, ηλιακής ενέργειας, ανεμογεννήτριες, τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες έχουν όμως και πολύ σοβαρές περιβαντολογικές επιπτώσεις. Ποια είναι η κατεύθυνση που δίνουμε εμείς. Τι θα κάνουμε, ας πούμε. Θα γεμίσει ο τόπος με αιωλικά πάρκα ή με ε, φωτοβολταϊκά συστήματα. Πράσινες οικονομίες είναι. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Ε, ένα δεύτερο ερώτημα για τις πόλεις για τις οποίες έγινε λόγος. Η βιολογική καθαρισμή ας πούμε ή το πρόβλημα της ανακύκλωσης των αποβλήτων που υπάρχουν προβλήματα σοβαρά και στην Ελλάδα από ό,τι ξέρω και στη Σλοβενία από ό,τι άκουγα τις προάλλες και σε πολλές άλλες χώρες. Αυτού του είδους τεχνολογίες θεωρούνται πράσινες ή όχι. Τρίτο ερώτημα. Είναι προφανές ότι μιλάμε είτε για νέους βιομηχανικούς κλάδους είτε για νέες τεχνολογίες. Αυτές βεβαίως μπορούν να ε, λυθούν σε επίπεδο περιφέρειας, όπως αναφέρθηκε πριν στην έκθεση που ψηφίσαμε, αλλά μιλάμε κυρίως για ε, ε, επιχειρήσεις και για κλάδους που προϋποθέτουν οικονομίες κλίμακας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί ούτε σε επίπεδο μιας περιφέρειας, ούτε στο επίπεδο μιας χώρας, εάν δεν εξασφαλιστούν όροι για μια μαζική παραγωγή και για μαζικές εξαγωγές. Αυτό πώς θα λυθεί. Θα πάμε πάλι στην ανταγωνιστικότητα και σε αυτά που έχουμε ζήσει με σοβαρά προβλήματα και στο θέμα της κάλυψης των αναγκών αλλά και, στην προκάλυ... και, στο να προκληθούν κρίσεις. Και τελειώνω. Νομίζω ότι εφόσον πρόκειται να αξιοποιηθούν ε, τα ε, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινωνικά ταμεία ή, ταμεία, ή κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής, πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και οι στόχοι της σύγκλησης. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάμε σε μια πράσινη οικονομία, παραδείγματο χάρη, η οποία να μην συνδέεται με την ανάγκη δημιουργίας μονάδων παραγωγής στην περιφέρεια, ώστε αντίστοιχα να μπορεί να καλυφθεί και το πρόβλημα της βιομηχανικής καθυστέρησης που έχουν πολλές περιφέρειες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Τσέλα. Äh, και εγώ ευχαριστώ και τις δύο συντηρήσει και την κυρία Βέσφαλ και την κυρία Σρότερ για τα όσα μας παρουσίασαν ε, σήμερα εδώ. Όταν κάνουμε λόγο για πολιτική συνοχή, όταν κάνουμε λόγο για περιφερειακή πολιτική, ένα από τα κύρια σημεία μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά την ε, προώθησή τους ήταν η υποστήριξη των περιφερειών έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και προκειμένου να δημιουργηθεί απασχόληση, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τώρα έγινε μια συζήτηση ότι η στρατηγική της Λισαβόνας 2000-2010 απέτυχε και ότι ο στόχος ε, του η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί η πιο δυναμική ε, βασισμένη στη γνώση οικονομία ε, και βασισμένη στην κοινοτομία Απέτυχε λοιπόν αυτή η πολιτική και ξαφνικά τι λέμε ότι έχουμε μια νέα πολιτική, πάλι έχουμε νέες προτεραιότητες, τι λέμε ότι είμαστε οι πρώτοι, οι καινοτόμοι σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών και θα έχουμε την πρωτιά σε αυτό το τομέα. Όλα αυτά είναι λίγο κοντόφθαλμα. Δηλαδή, ακόμα και στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας υπήρξαν κάποιους, κάποιοι τομείς ε, με επιτυχίες ε, και το έχουμε συζητήσει επανελειμμένα εδώ στην δική μας επιτροπή η πολιτική συνοχής ήταν ακριβώς ένα από αυτά τα στοιχεία με επιτυχία. Αν δούμε ε, το 2004 έως 2007 και την ένταξη τόσων πολλών νέων κρατών μελών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπιστώσουμε ότι υπήρξε και αλληλέγγυα υποστήριξη από την πλευρά των παλαιών κρατών μελών προκειμένου να ε, καταστεί δυνατή η προσχώρηση αυτών των νέων κρατών μελών και των περιφερειών τους. Και αυτό αποτελεί μια επιτυχία θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτές τις επιτυχίες μας σε ό,τι αφορά τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι σημαντικά και για τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί για αυτούς τους πολίτες χαράζουμε εμείς οι ε, πολιτικοί και για αυτούς τους πολίτες είναι σημαντικό να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους στο πλαίσιο μιας ε, διεθνούς οικονομικής κρίσης ή εν πάση περιπτώσει να ε, παραμείνουν ανοιχτές οι δυνατότητες για να ε, ε, παραμείνουν μέσα στην απασχόληση, μέσα στην αγορά εργασία. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να είναι σημείο προτεραιότητας όταν κάνουμε λόγο για την πολιτική μας σε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ τις δύο εισηγήτες. λοιπόν Ε, για το ότι αναφέρουν ίσως στην γνωμοδότηση της κυρίας Βεσφαλό, όχι τόσο πολύ, της κυρίας το πού βρίσκονται οι κινητήριες δυνάμεις, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ότι δηλαδή αυτά τα, τα κέντρα, αν θέλετε, είναι οι πόλη όπου μπορεί να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό. Και μέσα στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής ε, συνοχής θα πρέπει αυτή η διάσταση των πόλεων να ε, συνδεθεί η χρηματοδοτήσει σε επίπεδο ευρωπαϊκή πολιτική με τι περιφερειακέ ε, προσπάθειε. Γιατί είχαμε επιτυχίε στο παρελθόν σε αυτό το τομέα και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και να συνεχίσουμε να θυμόμαστε ότι η δημιουργία θέσεων εργασία σε απασχόληση αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία τη χάραξη περιφερειακής πολιτικής. Ευχαριστώ. Thank you very much. <coughs> was the last speaker. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Η κυρία Βέστφαλ. Συγγνώμη, κυρία Μανέσκου. Uh, ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας και να υπογραμμίσω δύο προτάσεις. Την υποστήριξη του πιλωτικού προγράμματος Έρασμος για την ανταλλαγή των τοπικών και περιφερειακών αντιπροσώπων και την κινητικότητά τους. Ελπίζω να δοθεί απαραίτητη ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλιστεί η συνέχιση αυτού του προγράμματος Έρασμος. Και πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών για να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Αυτή είναι η δεύτερη μου πρόταση. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, κυρία Βέστφαλ, θέλετε να δευτερολογήσετε, να σχολιάσετε τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Να, να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στο πλαίσιο της συζήτησης. Τα όσα εγώ άκουσα είναι ότι ε, δεν ήμουν τελείω εσφαλμένη στα όσα ανέφερα σε ό,τι αφορά την ε, περιφερειακή ανάπτυξη μέσα στο πολύ περιορισμένο ε, χώρο, στο κείμενο δηλαδή που είχα. Νομίζω πως όλοι κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή εράσμος από μία πλευρά και από την άλλη πλευρά ένταξη, ενσωμάτωση σε αυτή τη διαδικασία των τοπικών και περιφερειακών αντιπροσώπων και η προσέγγιση των επιχειρήσεων αποτελεί κάτι το σημαντικό εγώ προέρχομαι από αυτόν τον χώρο της ε, ε, πολιτική στο επίπεδο το τοπικό και από εκεί μετέβη ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική οπότε αντιλαμβάνομαι πολύ καλά το τι μπορούν να επιτύχουν οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντω, σε ό,τι αφορά την απασχόληση, το είπε μόλι τώρα ο κύριο Τσέλερ. Δηλαδή, βασικό στόχο είναι να διατηρηθούν οι θέσει εργασία και οι ποιοτικέ θέσει εργασία η κυρία Σότερ το ανέφερε επανειλημμένα, ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε ευνοϊκέ, σωστέ προποθέσει εργασία και όχι οποιασδήποτε θέσει εργασία. Και ε, αυτό αυτός είναι ένα τομέα ε, από του τομεί αρμοδιότητα τη Επιτροπή αποσχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εμεί θα πρέπει να εστιάσουμε στη δική μα διάσταση και ευχαριστώ εκ των προτέρων ε, του ε, συναδέλφου οι οποίοι θα συνεισφέρουν έτσι ώστε αυτή η γνωμοδότηση θα καταστεί ακόμα πιο σημαντική. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε. Ωραία, ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο. Μην ξεχνάτε συνάδελφοι ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει το μεσημέρι στις 4 Μαΐου. Θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση αυτή στις 22 Ιουνίου στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε κυρία Βέστφαρ και τους και οδησηγητές και περνάμε στο επόμενο σημείο, το 14, ανταλλαγή απόψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον ε, Διευθυντή Ρούντοφ Νίσλερ για ανταλλαγή απόψεων με θέμα τα πειραματικά και πιλωτικά προγράμματα που θεσπίστηκαν το 2009 μετά το αίτημα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ζητήσαμε πληροφορίες από τον Γενικό Διευθυντή πριν από ένα δίμηνο για την πρόοδο αυτών των σχεδίων και μάλιστα ο Γενικός Διευθυντής μας έστειλε επιστολή το Φεβρουάριο που σας διαβεβάσαμε και σήμερα καλωσορίζω στη συνεδρίασή μας τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ρέτζιο. Ελπίζω να έχουμε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων για τα πειραματικά αυτά σχέδια. Μάλιστα αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε την απόφασή μας για τον προϋπολογισμό του 2011 και θα αποφασίσουμε αν θα δώσουμε το πράσινο φως για τη συνέχεια αυτών των προγραμμάτων των πειραματικών σχεδίων και αυτό θα εξαρτηθεί και από τις δικές σας πληροφορίες Επίσης, ε, εξερευνούμε τη δυνατότητα και άλλων πιλωτικών προγραμμάτων. Θα είναι πολύ σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψεων για τις μελλοντικές μας αποφάσεις. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο και οργανώσατε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς δημοσιεύσαμε την έκθεση για την κατάσταση των προγραμμάτων το Φεβρουάριο. Αυτό που σας παρουσιάζω σήμερα μαζί με τον συνάδελφό μου και με τους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με τα πιλωτικά προγράμματα είναι κάποιες τελευταίες ενημερώσεις και εξελίξεις στα προγράμματα αυτά. μαζί με τα τέσσερα προγράμματα στα οποία θα αναφερθώ από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο. Υπάρχει και η συνεισφορά της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων που θα σας ε, μιλήσει για την υφαντουργία, για τα προγράμματα αυτά τα πιλωτικά στην υφαντουργία. Με τη βοήθεια του PowerPoint θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα διαφορετικά προγράμματα έτσι ώστε να μπορέσετε να τα κατανοήσετε πιο εύκολα. Καταρχάς, πανευρωπαϊκό συντονισμό των μεθόδων ε, ένταξης των Ρωμά. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα έχει σαν στόχο την υποστήριξη καινοτόμων αντιμετωπίσεων ε, κάποιων περίπλοκων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι Ρωμά. Προσπαθούμε ακριβώς να προωθήσουμε προγράμματα τα οποία να καλύπτουν πολλαπλές πτυχές των δυσκολιών της καθημερινότητας των Ρωμά. Υπάρχει μια σαφή σύνδεση αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων και της εξέλιξης των λειτουργικών προγραμμάτων, των κατεξοχήν προγραμμάτων μας δηλαδή, και η γνώση την οποία συλλέγουμε στα πλαίσια αυτών των πιλωτικών θα επηρεάσει και την ποιότητα της εφαρμογής των μέτρων υπέρ της συγκεκριμένης αυτής κοινότητας. Χρηματοδοτούμε τα προγράμματα αυτά, τα κυρίαρχα, από το Κοινωνικό και από το Περιφερειακό Ταμείο. Έχουμε έρθει σε επαφή με τους εμπλεκομένους Έγιναν δύο σεμινάρια στις 13 Μαρτίου και στις 26, 25 μάλλον Ιουνίου του 2009. Προσπαθήσαμε έτσι να καταλάβουμε καλά ποιες είναι οι καλύτερες ενέργειες τις οποίες θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε στα πλαίσια των πιλωτικών. Υπήρχαν τέσσερις βασικές προτεραιότητες τις οποίες καλύπτουν τα πιλωτικά προγράμματα. Ο πρώτος τομέας αφορά την εκπαίδευση και την φροντίδα των παιδιών σε προσχολική ηλικία. Η εκπαίδευση των παιδιών είναι κάτι το οποίο πρέπει να λειτουργήσει υπέρ αυτών των κοινοτήτων Προσπαθούμε να επηρεάσουμε τη ζωή των παιδιών αυτών, το ταχύτερο δυνατόν δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να προχωρήσουμε με καινοτόμες αντιλήψεις. Ο δεύτερος τομέας δράσης είναι η αυτοαπασχόληση και οι μικροπιστώσεις. Όπως γνωρίζετε η κοινότητα των Ρωμά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αγορά εργασίας είναι πολύ δύσκολο για έναν από την κοινότητα αυτή να γίνει υπάλληλο και γι' αυτό είναι πολύ καλύτερα να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, να αυτοαπασχοληθούν. Και γι' αυτό προτάθηκε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα υποστήριξης αυτής της αυτοαπασχόλησης μέσω και μικροδανείων, μικροπιστώσεων. Μια στήριξη ας πούμε 5.000 ευρώ μπορεί να βοηθήσει έναν Ρωμά να αγοράσει ένα μικρό αυτοκίνητο ή ένα όχημα γενικά και να μπορεί να κουβαλά τα προϊόντα του στις αγορές. Βασικός μας στόχος είναι να δώσουμε δηλαδή όθηση στην αυτοαπασχόληση. Το τρίτο θέμα είναι η πληροφόρηση και συνειδητοποίηση των προβλημάτων. Αυτό αφορά από τη μία την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τα συγκεκριμένα προβλήματα των Ρωμά και ενημέρωση για τις συνθήκες ζωής και κατοικίας. Και υπάρχουν και μέτρα που στοχεύουν στην ίδια την κοινότητα έτσι ώστε να υπάρξει μια αμοιβαία κατανόηση των προβλημάτων και το τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά, τα οποία μερικές φορές στο παρελθόν ήταν, ε, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερως αντιπαραγωγικά. Και τέταρτον, τα μέσα και οι μέθοδοι για την αξιολόγηση και τη συλλογή στοιχείων σαν βάση για, την, για τον καθορισμό πολιτικών δράσεων οι οποίες να εδράζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό θα μας βοηθήσει να συλλέξουμε προτάσεις οι οποίες στο μέλλον θα βελτιώσουν τις πολιτικές μας παρεμβάσεις στον τομέα αυτό. Η Γενική Διεύθυνση Regio είναι υπεύθυνη για το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Αποφασίσαμε όμως εμείς να δώσουμε προς τα έξω ένα μεγάλο κομμάτι της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών γιατί δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό για να φροντίσουμε μόνοι μας θεωρώντας ότι η γνώση και των ε, εταίρων μας θα μπορέσει να βοηθήσει τη δράση αυτή. Υπήρξε μια προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος για να προσκαλέσουμε εταίρους ιδιώτες στα προγράμματα αυτά και η διαδικασία αξιολόγησης ε, ολοκληρώθηκε το 2009 έγινε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι οργανώσεις οι οποίες επελέγησαν τους στείλαμε τον Μάρτιο του 2010 κάποια στοιχεία και βρισκόμαστε σε στάδιο διαπραγμάτευσης με τις οργανώσεις αυτές για κάποια θέματα πρακτικά, τεχνικά. Θα θέλαμε να μπορέσουμε να σας πούμε με ποιους θα συνεργαστούμε στο μέλλον. Καταρχάς με το Ταμείο Εκπαίδευσης των Ρωμά, για το θέμα της προσχολικής εκπαίδευσης. Στον τομέα της αυτοαπασχόλησης θα συνεργαστούμε με το Πολγκάρα Λαπιτβάνι και στην τρίτη περίπτωση με την Σπόλου International για την ενημέρωση και πληροφόρηση. 1,9 εκατομμύρια το πρώτο, 1,5 εκατομμύρια το δεύτερο και 0,9 εκατομμύρια το τρίτο. Το τέταρτο κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό για μας. Θα συνδυάσουμε τις δικές μας δυνατότητες με το Ταμείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και με την Διεθνή Τράπεζα, με το Παγκόσμια Τράπεζα. 400.000 δίδουμε στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και συνεργαζόμαστε με την Παγκόσμια Τράπεζα όπως είπα για να συλλέξουμε καλύτερα τα στοιχεία και να κάνουμε πιο προχωρημένες αξιολογήσεις. Αυτές οι δύο οργανώσεις, το Ταμείο του ΟΗΕ δηλαδή και η Παγκόσμια Τράπεζα, δραστηριοποιούνται στο θέμα της συμπερίληψης της κοινωνικής των Ρωμά εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν αρκετές χρήσιμες γνώσεις συλλέξει. Για το 2010 θα οργανώσουμε μία διάσκεψη το φθινόπωρο για τη συλλογή στοιχείων και την αξιολόγηση. Θα είδατε επίσης, εδώ βλέπετε και την επόμενη διαφάνεια, θα είδατε λοιπόν στο κτίριο Μπερλεμό μια πάρα πολύ μεγάλη αφίσα που δείχνει ακριβώς τις ανησυχίες που έχουμε και τη φροντίδα που δείχνουμε προς την κοινότητα αυτή. Είχε αναρτηθεί από την 4η Απριλίου μέχρι την 11η Απριλίου για την εορτή των Ρωμά η οποία ήταν η 8η Απριλίου. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιλωτικά προγράμματα, εκεί έχουμε προχωρήσει αρκετά και βρισκόμαστε σε συγκεκριμένη φάση εφαρμογής. Θα ήθελα να συνεχίσω τώρα με το δεύτερο πρόγραμμα τον έρασμο για τους τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες. when we started, ε, ε, ε, Όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτών των πιλωτικών δράσεων, είχαμε αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στα πλαίσια της κατανόησης του πώς θα ήταν σωστό να προχωρήσουμε. Είχαν απαιτηθεί ε, και πάρα πολλοί ανθρώπινοι πόροι και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ε, ε, επιβαρύνσεις πολλές πρακτικές εις βάρος αυτών οι οποίοι, για τους οποίους προορίζεται το πρόγραμμα, οι υποψήφοι δηλαδή για να μετακινηθούν ανάμεσα στις πόλεις της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να διασφαλίσουμε μια σωστή μεθοδολογία για την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων και να δείξουμε ότι οι μετακινήσεις αυτές, η κινητικότητα αυτή των τοπικών αρχόντων είναι χρήσιμη. Τα συγκεκριμένα, τα απτά αποτελέσματα αν θέλετε αυτών των ενεργειών δεν είναι εύκολο να τα διακρίνει κανείς. Και γι' αυτό έχουμε να κάνουμε περισσότερο με μια μακροπρόθεσμη διαδικασία διαμόρφωσης ικανοτήτων και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, τη μακροπρόθεσμη προοπτική δηλαδή. Για να υπάρξει ε, μια πιο ξεκάθαρη αντίληψη για τον τρόπο εξέλιξης των προγραμμάτων αυτών, ξεκινήσαμε μια μελέτη σε εισαγωγικά εφικτότητας. Ε, έναν εξωτερικό εργολάβο, το Εκοτέ και Κορίς, και αποφασίσαμε να ελέγξουμε δοκιμαστικά το ενδιαφέρον το οποίο θα, επιδεικνύει, θα ένα δείγμα εκλεγμένων τοπικών αρχόντων. Και διαλέξαμε επίσης να πάρουμε και σύμβουλες και στοιχεία για το τι είδους πρόγραμμα κινητικότητας θα ήταν το πιο χρήσιμο. Ζητήσαμε επίσης μια τελική έκθεση από τον εξωτερικό συνεργάτη μας μέχρι το τέλος του 2010. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση και τώρα έχουμε μια τέτοια έκθεση η οποία έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σε φάση διαπραγμάτευσης με τον εξωτερικό εργολάβο θα έλεγα. Εδώ σας δίνω κάποια από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης που δεν έχει ακόμα θα έλεγα καταλήξει σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε βάθη εμβάθυνση των στοιχείων αυτών. Πάντως μπορούμε να δούμε ότι πέραν του θέματος της διαθεσιμότητας σε επίπεδο χρόνου ενός τμήματος αυτής της ομάδας στόχου. Συζητήσαμε τα θέματα τα οικονομικά, τα θέματα της οικονομικής συμμετοχής και οικονομικής επιβάρυνσης και σε ποιους θα αναλογεί και κάποια άλλα θέματα όπως τα γλωσσικά εμπόδια, πώς να αντιμετωπίσουμε το ότι πάρα πολύ συχνά υπάρχουν περιορισμένες ικανότητες σε τοπικό επίπεδο των τοπικών αρχόντων να μπορέσουν να χρησιμοποιούν ξένες γλώσσες εύκολα. Είχαμε συζητήσεις επίσης για τη μορφή και τη διάρκεια την χρονική τέτοιου είδους ανταλλαγών που θα θέλαμε να προωθήσουμε. Συζητήσαμε επίσης για την σωστή μορφή την οποία θα πάρουν αυτές οι ανταλλαγές έτσι ώστε να έχουμε τα πλέον απτά αποτελέσματα. Έγινε μια γενική ανταλλαγή απόψεων ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα θέματα. Σε αυτή τη φάση βέβαια αυτό δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε κάποια γενικότερα προβλήματα. Πάντως ελέγξαμε και αντίστοιχα προγράμματα τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και του τι ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να δεσμεύσουμε εμείς για τη συγκεκριμένη ενέργεια. έχουμε πάντα υπόψη ότι όταν προτείνουμε τέτοιου είδους ε, μοντέλα, τέτοιου είδους πρότυπα, δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο αφορά μια αυστηρά θα την χαρακτήριζα περιηγητική δραστηριότητα. Αλλά έχουμε να κάνουμε με μια ανταλλαγή και μετακίνηση ανθρώπων οι οποίοι στοχεύουν στην πρόσκτηση γνώσης. Υπήρξαν επίσης 11 ομάδες εργασίας εμπλεκομένων τα λεγόμενα focus groups. Συναντήθηκαν εκεί τοπικοί και περιφερειακοί άρχοντες και ε, η ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα θετική. Οι πιθανοί υποψήφοι για τέτοιου είδους προγράμματα εξέφρασαν ένα ισχυρότατο ενδιαφέρον και θα πρέπει το ενδιαφέρον αυτό να το εξυπηρετήσουμε. Συζητήσαμε τα θέματα της διαθεσιμότητας χρόνου από πλευράς τους, όπως επίσης και ένα κάποιο, ένα κάποιο πρόγραμμα προπαρασκευής έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να συνεισφέρουν οικονομικά σε τέτοιου είδους προγράμματα. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ελέγξουμε. Τώρα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στο πρόγραμμα αυτό. Όπως γνωρίζετε θέλουμε να βοηθήσουμε και όπως ε, ακούσατε χτες αντιμετωπίζουμε την πρόταση αυτή Εράσμους δηλαδή με θετικό βλέμμα και συζητάμε τις δυνατότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται και ελέγχουμε επίσης τις δυνατότητες που μας δίνουν υπάρχοντα προγράμματα, προγράμματα συνεργασίας, για να δούμε αν θα μπορούσαμε μέσα σε αυτά τα προγράμματα να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί ήδη από τους τοπικούς άρχοντες. Είναι πρόωρο πάντως αυτό σε αυτή τη φάση να πω ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Να σας ζητήσω να μας δώσετε περισσότερο χρόνο για να εξετάσουμε τα μεθοδολογικά προβλήματα και να καταλήξουμε σε τελικές προτάσεις οι οποίες να είναι σωστά θεμελιωμένες και ε, με βάση τα δεδομένα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να κινητοποιήσουμε για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Για το επόμενο πειραματικό σχέδιο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ρόναλ Ντόλ για να σας παρουσιάσω αυτό το πρόγραμμα της ε, ενίσχυσης τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας μέσω της προώθησης περιφερειακής πολιτικής σε, γενικότερο, σε γενικότερη κλίμακα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Πρόεδρε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα όπως ξέρετε, αφορά ένα τομέα που σας ενδιαφέρει άμεσα ε, και ιδιαίτερα σας κύριε Πρόεδρε, μια και ήσασταν αρμόδια επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική. Και χάρη στους πόρους που κινητοποιήθηκαν μέσω του, του πιλωτικού προγράμματος, τα 2 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή για το 2009 και το 1,5 εκατομμύριο για το 2010 καταφέραμε να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα εν συντομία να σας υπενθυμίσω τους λόγους για τους οποίους θεσπίσαμε αυτό το πρόγραμμα. Ερμηνεύοντας την εντολή που μας ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά σε μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τρίτων χωρών ανάλογα με τις απαιτήσει τους για μεγαλύτερη συνεργασία και καλύτερη ενημέρωση για το πώς χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την περιφερειακή της πολιτική. Αυτό είναι ένα έντονο αίτημα από τις τρίτες χώρες. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάνω από 20 ετή πείρα, πολύ πλούσια πείρα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση περιφερειακών πολιτικών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Έτσι συμβάλλουμε και στην πρόθεση της εικόνας και την καλύτερη προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς. Μέσω της περιφερειακής πολιτικής έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να εξηγήσουμε σε τρίτες χώρες ποιες είναι οι προσφυλείς σε μας αξίες όπως είναι οι ανοιχτέ αγορές που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή πολιτική σε ό,τι αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού, τις δημόσιες προμήθειες, την αρχή της αηφόρου ανάπτυξης, του σεβασμού προ το περιβάλλον, της ισότητας των ευκαιριών. Είναι απαραίτητε προποθέσει που αποτελούν θεμέλιου λίθου της περιφερειακή πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μας ενδιαφέρει και στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες να προσπίσουμε αυτές τι αρχές. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του πιλωτικού προγράμματος για το 2009, θα μπορούσαμε να διαιρέσουμε το πρόγραμμα εργασία μα σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Καταρχήν, διοργάνωση σεμιναρίων και διασκέψεων με το θέμα αυτό. Δεύτερον, ανταλλαγή προγραμμάτων και ενδιαφερομένων σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες δράσεις οργάνωση μελετών και εκπόνηση μελετών και εκπόνηση κάποιων επικοινωνιακών εργαλείων. Δεν θέλω να δώσω έμφαση σε ένα πρόγραμμα εις βάρος άλλων. Θα σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση. 11 και 12 Μαΐου του 2009, για παράδειγμα, είχαμε την πρώτη διεθνή διάσκεψη για την περιφερειακή διακυβέρνηση σε σφαιρικό πλαίσιο με, στις Βρυξέλλες με 300 ε, συμμετέχοντες. Επίσης, τον Μάιο διοργανώσαμε πέρυσι και το σεμινάριο για την ΑΣΕΑΝ και τον Οκτώβριο είχαμε τις περιφερειακές Open Days. Επίσης, οργανώσαμε και μια διάσκεψη για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και ιδιαίτερα συνεργασίες για το χώρο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ε, ε, το χώρο ε, στην, στην Αφρική και το σεμινάριο αυτό έγινε στην Πουρκίνα Φάσο. Επίσης έγιναν ανταλλαγές αξιωματούχων και διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης. Ιδιαίτερα δραστηριοποιείται εδώ η Βραζιλία και είχαμε 40 εκπροσώπους της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε πώς εφαρμόζουμε την ε, περιφερειακή πολιτική, αν ασχολούμαστε με θέματα τομεακής και γεωγραφικής ε, εξάρτησης κτλ. Επίσης οργανώσαμε ανταλλαγές ε, αξιωματούχων και με την Κίνα και την Νοτιοανατολική Αγγλία για τα θέματα καινοτομία και τη διαχείριση των πόλων αριστείας με επίκεντρο την πόλη του Κέμπριτζ. Επίσης οργανώσαμε επίσκεψη εκπροσώπων έξι χωρών της Κεντρικής Αμερικής προς ισπανικές περιφέρειες και όπως ίσχυσε και για την επίσκεψη των Βραζιλιάνων ασχοληθήκαμε με θέματα εφαρμογής, μεθοδολογίας εφαρμογής για την περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης, ε, εξετάσαμε την δυνατότητα ιδρύσης ενός ε, υπερεθνικού αναπτυξιακού ταμείου για τις έξι χώρες και το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουν είναι το αναπτυξιακό, μοντέλο, ε, αναπτυξιακό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ταμείο Συνοχής. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που ενδιαφέρονται για παρόμοια προγράμματα. Το 2009 λοιπόν ε, εκπονήσαμε κάποιες μελέτες, ε, καταλήξαμε σε κάποιους όρους αναφοράς. Για παράδειγμα είχαμε μία μελέτη για την Ουκρανία, για τις προκλήσεις δύο συγκεκριμένων περιφερειών της Ουκρανίας. Επίσης, ε, ανασχολήθηκα με θέματα διασυνοριακά σε ό,τι αφορά το σύνδεσμο όμορων περιοχών της Λατινικής Αμερικής. Και μάλιστα φέτος θα υποβληθούν στο, ε, στο Εκουαδόρ τα πρώτα πορίσματα αυτής της ε, μελέτης. Έχουμε και ένα άλλο θέμα, για, μια άλλη μελέτη για το σύστημα συνεργασίας στο Μερκοσούρ, πάλι Λατινική Αμερική. Και εκεί θα γίνει και το θέμα της ε, εδαφικής αναθεώρησης της Βραζιλίας. Όλες αυτές οι δράσεις ξεκίνησαν, εγκαινιάστηκαν το 2009, τότε λήφθη σχετική απόφαση, αλλά περιμένουμε τα πορίσματά τους το 2010 και ίσως ε, και στις αρχές του 2011. Επίσης, όπως σας είπα, επεξεργαστήκαμε και κάποια επικοινωνιακά εργαλεία που θα τα προβάλλουμε στους εταίρους μας Ο τίτλος του είναι Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική, πηγή έμπνευση για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί βάλαμε ένα ερωτηματικό, γιατί είναι θέμα συμφωνιών και ανέβρεση συνένεσης. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τη δική μας, τους δικούς μας κανόνες διαχείρισης της περιφερειακής μας πολιτικής, ούτε θέλουμε να υπαγορεύσουμε ή να καθοδηγήσουμε στις υπόλοιπες χώρες εκδίδωσε ένα εγχειρίδιο περιφερειακής πολιτικής, όλα είναι θέμα συνένεση. Πάντω ο διάλογος αυτός σε αυτά τα θέματα είναι πολύ χρήσιμο. Για το 2010 συνεχίζεται η προσπάθεια και χρησιμοποίησα μερικούς από τους εναπομείνοντες πόρους του 2009, κάποια κονδύλια που είχαν μείνει αναξιοποίητα για φέτο προβλέπονται αρκετές δράσεις. Για παράδειγμα, υποστηρίξαμε την διοργάνωση των ε, Open Days στη Βραζιλία, κατά το πρότυπο των Open Days στις Βρυξέλλες, με θέμα πάλι την αναπτυξιακή πολιτική. Θα διοργανώσουμε σεμινάρια για αξιωματούχους της Βραζιλιάνικης Διοίκησης για τεχνικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής, όπως ε, μέθοδοι αξιολόγησης, ε, έλεγχος ε, δημοσιονομικός και χρηματοπιστωτικός, ε, συνδρομή σε θέματα ανταλλαγή πληροφοριών. Συνεργαζόμαστε και με την Κίνα για μια διεθνή έκθεση που θα γίνει στη Σανγκάη για θέματα περιφερειακής πολιτικής. Και η Αργεντινή αρχίζει και να αναδύεται ως χώρα που επιθυμεί βαθύτερο διάλογο με τον ΩΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε το έργο μας με την Ουκρανία και η Νότια Αφρική επίση ε, υπέβαλε έτοιμα για συνδρομή, το ίδιο και η Αυστραλία για θέματα περιφερειακά. Βέβαια, επίκεντρο τη προσοχή μα είναι οι τέσσερι χώρε που ήδη έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μνημόνια Κατανόηση. Την Κίνα, τη Ρωσία δηλαδή, τη Βραζιλία και την Ουκρανία. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις ad hoc ε, αιτήσει και άλλων περιοχών ανάλογα με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Βέβαια, είναι απρόβλεπτες οι εξελίξεις και δεν μπορούμε να ξέρουμε κάθε μήνα τι αιτήσεις θα υποβάλλονται. Είναι και θέμα διοικητικής συνεργασίας. Το 2009, για παράδειγμα, δεν είχαμε ιδιαίτερη συνεργασία με τη Ρωσία, κάτι που ανατράπηκε το 2010, που έχουμε μεγάλη δραστηριοποίηση. Το αντίστροφο συνέβη με την Κίνα. Το 2009 είχαμε πολύ έντονη συνεργασία, ενώ φέτος ε, είναι πιο χαλαρή. Πάντως σίγουρα τα αιτήματα ξεπερνούν τις δυνατότητές μας. Και πολλές διοικήσεις ανά τον κόσμο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το μοντέλο ανακατανομής που αποκαλούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτικής Συνοχής. Και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, αν ήταν μόνη της την προσπάθεια αυτή, θα είχε τεράστιες δυσκολίες να ανταποκριθεί σε, στην πληθώρα αυτή ετοιμάτων. Αλλά χάρη στα πιλωτικά προγράμματα είχαμε μια πολύτιμη υποστήριξη και έτσι καταφέραμε να έχουμε πολύ καινοτόμε ανταλλαγέ και συνεργασίε που θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν χωρί τη συνδρομή αυτού του προγράμματο. Γι' αυτό και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη αυτή και το λέω αυτό και παρουσία τη κυρία Χιούμπνερ που είναι και η, η πρόεδρος αλλά και παρουσία του κυρίου Βανίλη Ρόι που είχαμε πολύ στενή συνεργασία για την υλοποίηση του προγράμματο αυτού του τελευταίου 18 μήνα. Και μάλιστα όλοι όσοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολούμαστε με το θέμα αυτό είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία να κάνουμε την αυτοκριτική μας για θέματα περιφερειακής πολιτικής. Γιατί πρώτα αυτό θα πρέπει να διαρωτηθούμε. Τι κάνουμε εμείς στην ε, περιφερειακή πολιτική για να μπορέσουμε στη συνέχεια να το εξηγήσουμε και να γίνει κατανοητό και στις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ρόνι. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το τέταρτο πιλωτικό πρόγραμμα, την τέταρτη πιλωτική δράση που ονομάζεται προπαρασκευαστική δράση για την πρόθεση ε, καλύτερου περιβάλλοντος, πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις μικροπιστώσεις. Στην προπαρασκευαστική αυτή δράση προβλέπονται 7 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα κονδύλια που ε, έδωσε η ΕΤΕ για το Jasmine. Το τεχνικό μέσο δηλαδή για την πρόθεση ε, δυναμικού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν μικροπιστώσεις και που δεν είναι τράπεζες. Και προβλέπονται και κάποιες επιδοτήσεις ε, του ΑΕΦ που θα προσθεθούν. Έτσι θα συμβάλλουμε και εμείς στις προσπάθειες προαγωγής των μικροπιστώσεων. Αυτά τα 7 εκατομμύρια τα χωρίσαμε σε δύο δόσεις θα δοθούν στο EIF που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δράσεων και του Jasmine και της ΕΤΕ και μάλιστα οι διευκολύνσεις προόδου θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη διαχείριση. Το 2009 δώσαμε επιδότηση 4 εκατομμύρια και το 2010 θα χρησιμοποιηθούν τα 3 εκατομμύρια που απομένουν από το συνολικό ποσό των 7 εκατομμύρια. Όταν έχουμε τέτοιες συμφωνίες επιδοτήσεων με το Ταμείο Επενδύσεων, το Ταμείο Επενδύσεων θα προσθέσει ένα συμπληρωματικό κονδύλιο που θα ανέλθει σε 250.000 ευρώ. 250.000 ευρώ. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης που πρικοδοτείται με 7 εκατομμύρια. Καταρχήν θα δοθεί ένα βασικό κεφάλαιο για τα ιδρύματα αυτά που χορηγούν μικροπιστώσεις και που δεν είναι τράπεζες. Στόχος μας είναι πέντε κυρίως τέτοιοι πάροχοι μικροπιστώσεων για το 2009 και τρεις με τέσσερις τέτοιοι πάροχοι για το 2010. Οπότε συνολικά οι πάροχοι που θα εμπέσουν στο πρόγραμμα είναι 8 με 9. Και 900.000 ευρώ είναι ο μέσος όρος συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα και έναν εμπορικό χαρακτήρα σε μεσοπρόθεσμη πρόπτικη για τα αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παροχής μικροπιστώσεων. Τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επενδυθούν σε μία τετραετία μετά την ε, μεταβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το μέσο αυτό διευκόλυνσης θα ολοκληρωθεί το αργότερο τέλη Δεκεμβρίου του 2017. Για τη διαχείριση των δράσεων αυτών προβλέπεται ένα κόστος διαχείρισης ε, που θα ανέλθει στο 7% του ποσού. Το 7% όμως θα καλύπτει ολόκληρη την περίοδο, μέχρι το 2017. Άρα δεν είναι υπέρογκο το ποσό της διαχείρισης. Τι προβλέπετε για το 2010. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία των διαφόρων δραστηριοτήτων στα θέματα μικροπιστώσεων, προκειμένου να ενδυναμώσουμε την αποτελεσματικότητά τους και να διαμορφώσουμε κάποιες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων φορέων. Μάλιστα θα έχουμε και τη συμβολή του Progress. Η αρχική πρόταση στα πλαίσια του Jasmine και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εμπλουτίστηκε με μια νέα διάσταση. Δεν έχουμε μόνο δηλαδή τη συνεισφορά για το capacity building, και την δυνατότητα δανεισμού 40 εκατομμυρίων όπως προβλεπόταν αρχικά. Τώρα έχουμε και μια νέα διάσταση και μάλιστα η ΕΤΕ θα ενισχύσει την συμβολή της. Γι' αυτό και σε συνεργασία με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Επασχόλησης και ΕΚΦΙΝ που ασχολείται με το συντονισμό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Αυτά για το 2010. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε το κατάλληλο μοντέλο για να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες των μικροπιστώσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με μεσοπρόθεσμη προοπτική. Χωρίς να αφισβητούμε φυσικά την αφετηρία του Τζάσμιν και την συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τις πρώτες τέσσερις πιλωτικές δράσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Περίεργο. Και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του συναδέλφου, γιατί χθε μίλησα, είχα τηλεφωνική συνομιλία με κάποιον από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και με διαβεβαίωσαν ότι θα, θα υπήρχε εκπρόσωπο στη σημερινή συνεδρίαση. Λυπάμαι γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες ενδεχομένως. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε 25 μόνο λεπτά για τη συζήτηση μας. Ο Λομπέρ Βασινστελό, πρώτος ομιλητής και ο πρωτεργάτης αν θέλετε αυτού του Global Approach είναι πολύ καλή αυτή η ενημέρωση για, την, ε, για το γεγονό ότι την ε, ακούμε τώρα ε, στην Επιτροπή μας, ούτω ώστε να γνωρίζουμε το πού βρισκόμαστε αλλά και το προς το πού κατευθυνόμαστε. Το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι τα πιλωτικά προγράμματα αποτελούν μια δυνατότητα για το Κοινοβούλιο να καταστήσει δυνατά επιπρόσθετα σημαντικά στοιχεία τα οποία τελικά θα, αργότερα θα αποτελέσουν μια αυτόνομη ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού της Ένωσης. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί δοκιμάζουμε κάποια πράγματα ούτως ώστε αργότερα να τα καταστήσουμε ένα σταθερό αν θέλετε στοιχείο των ε, τρέχοντων ε, προτεραιοτήτων. Ε, χρειαζόμαστε δύο-τρία χρόνια ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχει κάτι έχει πετύχει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτά τα στοιχεία μας δίνουν ε, κάποια, κάποιες επιπρόσθετες μονάδες αν θέλετε, αλλά από εκεί και μετά δεν θα πρέπει να αναμένουμε ε, πάρα πολύ ε, ούτω ώστε να ενσωματώσουμε αυτά τα, αυτές τις μονάδες, αυτά τα στοιχεία στις κανονικές ε, προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και αυτό επαφείται και σε εσά, Πρόεδρε, δηλαδή το πώς θα κάνουμε μια συνολική, αν θέλετε, πρόταση από την πλευρά της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του 2011, 2012 και πιο μετά μετά. Σε ό,τι αφορά τις την ε, ενημέρωση, επιτρέψουν να κάνουν κάποια πολύ επιγραμματικά σχόλια, να μην επισέλθω σε λεπτομέρειε. Καταρχήν, στο πρώτο πρόγραμμα για του ΡΟΜ. Ε, είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε τώρα κάποιε προτάσει ε, και γνωρίζω πω η σοσιαλιστική ομάδα είχε το στο έναυσμα για αυτή την ιδέα. Οπότε καλό θα ήταν να υπάρχει μια καλή επικοινωνία με όσους είχαν κάνει την αρχή εδώ, είχαν κάνει τις αρχικές προτάσεις ούτω ώστε να βλέπουμε κατά πόσο σημειώνεται πρόοδο ή όχι. Ε, θεωρώ πως υπάρχει πρόοδο και είναι δύσκολο να φτάσει κανείς στη βάση αν θέλετε των ανθρώπων αυτών και να καταστήσει δυνατή μια αλλαγή μακροπρόθεσμα. Ε, θεωρώ πάντως πως υπάρχει αλλαγή. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το υποστηρίξουμε στο μέλλον αυτό το πρόγραμμα και το πώς μπορεί να ενσωματωθεί ε, στην ε, κανονική αν θέλετε, πολιτική. Μετά, το πολιτικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το αρέσμος. Προτάθηκε από τους φιλελεύθερους ε, ήδη ή μάλλον τέθηκε επιτάπητος ότι δεν τρέχει όπως θα θέλαμε. Γιατί αν βλέπαμε κανονικά τα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι είναι δύσκολο να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που θέλαμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου είναι να υπάρξει μια νέα όθηση με αυτή τη νέα προσέγγιση, ούτω ώστε οι άνθρωποι στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και θεωρήσαμε ε, πως κάποιες από τις γενικές ε, από τους συνολικού φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή των Περιφερειών, να αναλάβουν έναν ηγετικό ρόλο όπως για παράδειγμα τα μικροδάνα, τα macro credits. Αλλά είναι ε, δύσκολο μετά γιατί υπάρχουν χιλιάδες ερωτήσεις που απευθύνονται προς την ε, Επιτροπή πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο, πώς θα χρηματοδοτηθεί και ούτω καθεξής και τελικά στο τέλος δεν ε, έχει γίνει τίποτα. Χρειαζόμαστε συνήθως δύο χρόνια για μια τέτοια πρωτοβουλία. Δεν έτρεξε το πρόγραμμα όπως ε, είχαμε προβλέψει. Ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Ε, για να έχουμε ένα κανονισμό ή κάτι αντίστοιχο το οποίο να διασφαλίζει ότι θα δαπανώνται με τον τρόπο που θέλουμε τα κονδύλια αυτά. Αλλά πραγματικά έχω ανησυχίες για το αν θα συνεχίσουμε έτσι με αυτό το πρόγραμμα, γιατί χάνουμε μια ευκαιρία. Μετά, σε ό,τι αφορά την ε, ενίσχυση της ε, τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας, είναι θετικά τα όσα βλέπουμε εκεί. Έχουμε ήδη, είχαμε ήδη επικοινωνία στο παρελθόν μεταξύ μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια συνεργασία, δεν αναφέρεται μόνο στις ε, κλιματικές μεταβολές ή στις διαπραγματεύσεις στο επίπεδο του ΟΠΟΕ. Υπάρχουν πολλά πέραν αυτών. για να δοθεί η δυνατότητα της καλής ανάπτυξης μέσω μιας συνολικής ε, προσέγγισης ε, και στο επίπεδο των περιφερειών και στο επίπεδο των πόλων. Άρα λοιπόν, εάν ε, θέλουμε να επιτύχουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό το τάβμα, το πούμε έτσι, με αυτή τη μεταμόρφωση την οποία επιτύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να οπισθοχωρήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή με τον τρόπο, με την ταχύτητα την οποία αναπτύξαμε, χωρίς δηλαδή να κάνουμε βήματα προ τα πίσω. Και ε, είπατε επανειλημμένα ότι έχετε ε, πολύ καλή συνεργασία ε, στην Επιτροπή, με, την, ε, με τον ΩΣΑ και ούτω καθεξής, αλλά θα ήθελα να ξέρω ε, ποιο είναι το επίπεδο της συνεργασίας με τα μέλη του Κοινοβουλίου. Αντιλαμβάνομαι την πρόθεσή σας, ε, το θετική σας πρόθεση, αλλά όταν υπάρχουν ε, σημαντικές συνεδριάσεις από την πλευρά σας, να αποστέλλετε στις πολιτικές ομάδες ή δεν ξέρω με ποιον τρόπο να μας ενημερώνετε. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, να μας δίνετε τη δυνατότητα να δίνουμε και εμείς την αμυγός ευρωπαϊκή, αν θέλετε, διάσταση ως ελευθερία αντιπροσωπή από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θεωρώ πως ε, το λόγο σημείο θα πρέπει να αποτελέσει μια κανονική γραμμή του προπολογισμού μακροπρόθεσμα. Δεν χρειάζεται να το κάνει δηλαδή μόνο αυτό το τμήμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ένα ρεαλιστικό ζήτημα εδώ. Και εγώ ήμουνα πρόεδρο τη Ένωση για τι Συνοριακέ ε, Περιοχέ και έχουμε εδώ το πρόγραμμα Interreg και αυτέ τι νέε περιοχέ των Πυρενέων και αλλού οι οποίε δεν υπάρχουν, για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική. Και υπάρχουν πολλέ δυνατότητε οι οποίε χάνονται επιτόπια σε ό,τι αφορά την διαδοχωματική περιθάλψη, το εμπορίο και ούτω Και εκείνη η Λατινική Αμερική μα ρωτάει τώρα ε, πόσο μπορούμε εμεί, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο να ε, διασφαλίζουμε αυτήν την διασυνοριακό αν θέλετε χαρακτήρα διαπεριφερειακή ε, οικονομική συνεργασία γιατί δεν έχουμε ένα σύστημα με αυτό που έχουμε τώρα. Μπορούμε λοιπόν να παρουσιάσουμε ακριβώ το ότι έχουμε κάνει εμεί χωρί να υποδεικνύουμε στον υπόλοιπο κόσμο το πώς, ποιο μοντέλο θα, ποια προσέγγιση θα χρησιμοποιήσουν. Χωρί δηλαδή να θέλουμε να πούμε ότι οι δικέ μα ιδέε ή τα δικά μα κριτήρια είναι τα μόνα που μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο μια τέτοια συνεργασία. Σε ό,τι αφορά μικροδάνεια. πραγματικά είναι μια περίπτωση όπου μικρές ιδέες μπορούν να έχουν μεγάλο αποτέλεσμα και νομίζω πως μπορούμε να το επιτύχουμε στη συνεργασία με άλλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σωστό κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει κανείς να κάνει κάτι μόνος του. Θα πρέπει να το οργανώνει σωστά και μετά συμμετέχουμε όλοι. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα δεν θα πρέπει να σταματάει αν όλοι είναι ευχαριστημένοι. Οπότε καλώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σκεφτούν το κατά πόσο μπορούν να οργανώσουν καλύτερα μια τέτοια πρωτοβουλία. Ας μην προσπαθεί δηλαδή μόνη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιλύσει όλα τα προβλήματα, δηλαδή να λαμβάνει την καθοδήγηση, τη διαχείριση και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την ενημέρωση και θα θέλαμε η ε, γραμματεία εδώ να παρέσει αντίστοιχη ενημέρωση ό,τι αφορά την αξιολόγηση και ούτω καθεξής και ε, να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και εμείς από την πλευρά μας ε, για την περίοδο 2011-2013 για νέες ιδέες και υπάρχουν κάποιες νέες ιδέες ούτως ώστε η κατάσταση της πόλης, η διάσταση των πόλεων να τεθεί εδώ ως προτεραιότητα. Εν πάση περιπτώσει, ας σκεφτούμε κάποιες ε, δυνατότητες, κάποιες ιδέες. Oui, Αυτές οι τέσσερις πρωτοβουλίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα ποιότητας παρουσίασης για τους Ρώμα σαν παράδειγμα. Αυτό το οποίο προβλέπετε είναι θετικό και ελπίζω να προσφέρει αποτελέσματα. Η απογοήτευση όμως είναι μεγάλη για το έρασμος που αφορά τους ε, ε, τοπικούς άρχοντες. Βλέπουμε ότι δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να βρούμε λύσεις συγκεκριμένες για ένα πρόγραμμα το οποίο ε, σημαίνει πολλά για μας, γιατί ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη. Λοιπόν, δεν είναι παραγωγικό το να κουβαλάει κανείς τους Πορτογάλους στη Φιλανδία χωρίς να έχουν τη δυνατότητα μετάφρασης προφανώς. Μήπως μπορούμε να πάμε ανάποδα, δηλαδή να προτείνουμε μέσα από συγκεκριμένες προκηρύξεις ενδιαφέροντος, κάποιοι δήμοι, κάποιες κοινότητες που έχουν αποδείξει ότι έχουν δυνατότητες σε κρίσιμους τομείς σχετικούς με την κινητικότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την προστασία της βιοπικιλότητας, γενικά τομείς οι οποίοι πήγαν καλά μέχρι τώρα να γίνουν ε, πόλεις υποδοχής θα έλεγα Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις συγκεκριμένες κοινότητες που έχουν ε, πρακτικές οι οποίες είναι χρήσιμες με κάποιες θεματολογίες οι οποίες να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σύνολο των Ευρωπαίων. Θα πρέπει λοιπόν οι πιο προχωρημένες αν θέλετε κοινότητες να χρησιμοποιηθούν πρώτα για την εξυπηρέτηση και των υπολείπων. Για το τρίτο θέμα. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα. Για τις μικροπιστώσεις. Εμείς περιμένουμε πολλά από αυτά τα οποία γίνονται. Ελπίζω να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και γρήγορα. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που περιμένουν το λόγο. Όχι. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θα μου επιτρέψετε να θέσω. Νομίζω ότι ένα από τα πιο βασικά θέματα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τα πιλωτικά αυτά προγράμματα να μην παραμείνουν ε, προγράμματα εφάπαξ θα έλεγα. το θέμα της αηφορίας και το θέμα του το τι πραγματικά περιμένουμε από το σύστημα είναι πολύ σημαντικό για μας. Γι' αυτό το πρόβλημα ε, σχετικά με το Εράσμους είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για μας. Συζητήσαμε το θέμα αυτό και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο γιατί πιστεύουμε ότι ο ρόλος αυτών των επιπέδων διακυβέρνησης στην Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς. Το να βελτιώνεται η ποιότητα της διακυβέρνησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι επίσης πολύ θετικό. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται να βελτιώσουν την ποιότητα της δουλειάς τους και ακριβώς αυτό το Εράσμος δημιουργήθηκε έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο θα έλεγα στην απόδοση των τοπικών αυτών μορφών διακυβέρνησης και να βελτιώσουμε εν πάση περιπτώσει την απόδοσή τους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε τώρα. Συνειδητοποιώ όλα τα προβλήματα που υπάρχουν ε, προφανώς δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λειτουργεί ε, σαν γραφείο ταξιδίων, αυτό είναι σαφές. Αλλά αυτό το οποίο είπατε, αν κατάλαβα καλά, αντιμετωπίζετε τη δυνατότητα να εντάξετε το πρόγραμμα αυτό σε ένα από τα υπάρχοντα προγράμματα, τα οποία είναι υπό εξέλιξη, όπως το Urban σαν παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Το να θεωρήσει κανείς ότι το εράσμος είναι μια προτεραιότητα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει να ενταχθεί στα πλαίσια των ε, πιο ε, συνηθισμένων και δρεωμένων πολιτικών που ακολουθούμε. Συζητάμε στα πλαίσια της Επιτροπής μας και το δημοσιονομικό κανονισμό που θα δημιουργήσει το πλαίσιο για τις μελλοντικές πολιτικές μας. Ξέρω πόσο δύσκολο θα είναι να υπάρξουν αλλαγές αργότερα στο δημοσιονομικό κανονισμό. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια της συζήτησης αυτής ίσως θα πρέπει να βρούμε και κάποιες δυνατότητες έτσι ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να μην χρειάζονται τόσα χρόνια έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα με όλα αυτά τα πιλωτικά προγράμματα γιατί επαναλαμβάνω χάνουμε πάρα πολύ χρόνο λόγω των ε, κανόνων που είναι σε ισχύ. Θα πρέπει να προσπαθήσετε κι εσείς να δείτε τι μπορεί να γίνει και στα πλαίσια της πολιτικής για τις πόλεις, γιατί είναι κάτι που συνδέεται άμεσα με το Εράσμους αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι κάτι το οποίο πολύ σημαντικό για μας και αυτό το είπε ο Λαμπέρ και για κάποιους άλλους που είναι απόντες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τον οποίο προωθούμε τα προγράμματα αυτά. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό ποσοτικά εννοώ και οι άνθρωποι που απασχολούνται με ορισμένα θέματα στην Επιτροπή αναγκάζονται να αναλαμβάνουν συνεχώς και περισσότερα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το λάβουμε υπόψη μας όταν προωθούμε τέτοιου είδους νέες κατά τα άλλα πρωτοβουλίες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τα πιλωτικά προγράμματα να συνειδητοποιήσουμε το βάρος που αντιπροσωπεύουν έτσι ώστε να μην απαιτούνται τόσα χρόνια για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να καταστήσουμε τις πρωτοβουλίες αυτές τις οποίες αναλαμβάνουμε εφικτές. Και τέλος, κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού, είναι το πώς θα εμφαρίνουμε κάπως τα πράγματα, θα τα διευκολύνουμε μέσω της αύξησης των πόρων που είναι διαθέσιμη για να βελτιωθεί και η συνεργασία ανάμεσα στις γενικές διευθύνσεις. Για τους Ρωμά, νομίζω ότι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει στο μέλλον να γίνει ένα εδρεωμένο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να γίνουν προτεραιότητα. Θα πρέπει να αντακαταστήσουμε mainstream προγράμματα στο μέλλον. Ο τρόπος που θα ασχοληθούμε με την ε, μειονότητα των Ρωμά στο μέλλον νομίζω είναι καθοριστικός. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σχόλιά μου και θα ήθελα να ζητήσω από όλους να σκεφτούμε περισσότερο την δυνατότητα να εξελιχθεί έτσι το πρόγραμμα αυτό Εράσμους, έτσι ώστε να δούμε τα αποτελέσματά του γρήγορα. Συγγνώμη που σας καθυστερώ, αλλά είναι... άκουσα μετά, μετά τη συζήτηση που είχαμε για το Έρασμος Πιστεύω ότι ειδικά στην Επιτροπή μας θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τις νέες πρωτοβουλίες. Για, την, για τον Τζέσικα, για παράδειγμα. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και οι τοπικές αρχές ε, όταν συνάντησαν την ΕΤΕ και διαπίστωσαν πόσο ε, δαπανηρό είναι το πρόγραμμα, είπαν ωραίο μεν, αλλά άχρηστο. Τώρα η ΕΤΕ άλλαξε κάπως την πολιτική της και στην Πολωνία πρότεινε ένα ελάχιστο επίπεδο που είναι απαράδεκτο για, για μας. Και όταν υποβάλλουμε μία νέα ιδέα που είναι ενδιαφέρουσα θα πρέπει να είναι και εφικτή και απλή και εύληπτη. Αλλιώς θα επιβεβαιώσουμε το φόβο των πολιτών είναι τόσο περίπλοκη η ευρωπαϊκή πολιτική που είναι αδύνατο κανείς να τη χρησιμοποιήσει. Το έρασμος ήταν απλούστατη ιδέα. Ο την πρότεινε ως ένα πλούστατο ζήτημα. Οι τοπικές ε, αρχές να μπορούν να διδαχθούν ημένα από τους ΔΕ και στο Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών EuroCities χρησιμοποιούσαν ε, τέτοιες ε, δραστηριότητες χρόνια ολόκληρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με τις γλώσσες ούτε με τη διοργάνωση. Γιατί ούτως ή άλλως οι τοπικοί σύνδεσμοι τα είχαν, είχαν κάνει τέτοιες διοργανώσεις. Και δεν υπάρχει πρόβλημα με τη γλώσσα, γιατί φυσικά μόνο όσοι γνωρίζουν γλώσσες ταξιδεύουν. Αλλιώς χρειάζονται και διερμηνία, κάτι που αυξάνει το κόστος του προγράμματος. Θυμάμαι πριν την ένταξη, όταν διαπραγματευόμασταν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε τον Ζαν Σαρλέγκ και εμείς ε, προσπαθούσαμε να εξετάσουμε πώς θα εντάξουμε το Eco Μετά από μήνες, πολλοί μήνες διαπραγματεύσεις, τελικά την πλήρη διοργάνωση την ανέλαβε το CMR, δηλαδή το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών. Τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκούσε μόνο την εποπτεία. Και είναι σημαντικό για τα νέα δοκιμαστικά και πυλαματικά προγράμματα. Αν προτείνουμε κάτι, θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλιώ θα, θα περάσουμε στην διακυβερνητική Ευρώπη, κάτι που έκανε η Λισαβόνα. Αλλά εμεί θέλουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη και μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να επιφορτίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μικροπρογράμματα 2 εκατομμυρίων και μετά από δύο χρόνια να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι περίπλοκη η διαχείρισή του. Δηλαδή να ξοδέψουμε ένα από τα 2 εκατομμύρια για να ε, διαπιστώσουμε τελικά ότι είναι περίπλοκο το πρόγραμμα. Δώστε εμά το 1 εκατομμύριο, θα σα το πούμε σε μια εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να περάσει ένα χρόνο. Και αυτή είναι η παγίδα των ε, προγραμμάτων μικρής εμβέλειας. Και αν πρόκειται για μια δοκιμαστική δράση, αν είναι μια πειραματική δράση, ένα δοκιμαστικό ή πιλωτικό πρόγραμμα, θα πρέπει αμέσως να το προτείνουμε. Σε ένα από τους βασικούς φορείς, το CMR, CPRM, έχουν προσωπικό και δυνατότητα να το διοργανώσουν και θα μας βγει και φτηνά. Ακόμη και η Επιτροπή Περιφερειών μπορεί να αναλάβει τέτοια μικρή εμβέλειας σχέδια. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σωστό μάθημα που θα πρέπει να διδαχθούμε. Δεν επικρίνω την Επιτροπή. Γιατί για να την αναλάβετε σε αυτή τη δουλειά θα πρέπει να κάνετε αξιολόγηση, εκτίμηση εξάντε, αξιολόγηση εξπόστ, ανάλυση σκοπιμότητας, ανάλυση βιωσιμότητας και έτσι περιπλέκονται τα πράγματα και τελικά δεν οδηγούμε πουθενά. Είτε θα έχουμε δοκιμαστικό πρόγραμμα και πιλωτικό πρόγραμμα και μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας σε τοπικό επίπεδο πολύ καλά. Γιατί δεν είναι καλή και στις 20 Μαΐου θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα βέλτισης πρακτικής. Και έχουμε μερικά τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη. Γιατί να μην στέλνουμε τα κονδύλια αυτά κόσμο εκεί, χωρίς προκηρύξη επίσημης διαγωνισμών και αναλύσεις επί αναλύσεων. Απλώς να περάσουμε στη δράση και όχι οι λόγια. Γιατί να μιλούμε για δύο ώρες για ένα μικρό πρόγραμμα 2 εκατομμυρίων, φανταστείτε θα γίνει μετά από ένα χρόνο. Θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Ας μείνουμε απλοί και ας μην επιφορτίζουμε με τέτοιες μικρολεπτομέρειες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό στο μέλλον ως καθοδηγητικό πρόγραμμα. Εσείς είστε αρμόδιοι για δισεκατομμύρια. Τώρα θα συζητούμε τέτοια ψυχία, μικροπρογράμματα 2 εκατομμυρίων. Ευχαριστώ Γιάννη και πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη αυτό όταν θα εξετάσουμε κανονισμούς που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με τρόπο που δεν θα προκαλέσει τους κεραυνούς του ελεκτικού συνεδρίου που θα ζητήσει ανάκτηση των κονδυλίων ή επαναφορά και στις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές όλοι θα ρίναμε πρώτα απ' όλα της Ευρωπαϊ... και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ίδιο τις περιφέρειες να δείξουν καινοτομία. Αλλά μετά είχαμε το λεπτικό συνέδριο που τα αφισβήτησε όλα αυτά. Προσοχή λοιπόν στους κανονισμούς. Ίσως εκεί θα πρέπει να πούμε ότι τα πιλωτικά προγράμματα διέπονται από ειδικού κανόνες που μας επιτρέπουν να παρεκκλίνουμε από τους γενικούς κανόνες και τις γενικές αρχές περί προκήρυξης διαγωνισμών κτλ. Ναι. Μα αυτή είναι η απλούστευση που ζητούμε. Αλλά θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιληφθεί ότι ο δημοσιονομικό κανονισμό που θα υιοθετηθεί τέλη Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα θέσει το πλαίσιο για την επόμενη πενταετία ή επταετία μπορεί να σκοτώσει στα σπάργανα όλες τις καλές μας ιδέες και προτάσεις. Θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα, ένα παραθυράκι για όλα αυτά τα πειραματικά προγράμματα και τις δοκιμαστικές δράσεις, ώστε να είμαστε πραγματικά άμεση δράση και ελπίζω να χρησιμοποιηθεί αυτή η συζήτηση για να φανεί και ο νομοπαρασκευαστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει έχει τρία με πέντε λεπτά το πολύ. Κυρία Πρόεδρε, να κάνω κάποιε επιλεκτικέ ε, παρατηρησει ε, σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν. Όταν ο κ. Ολμπριχτ έκανε λόγο ε, για τις δυσκολίε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση τέτοιων μικρότερων εργών, είχε απόλυτο δίκιο, αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε ένα πράγμα εδώ. Πριν από όχι πολύ καιρό, είχε ληφθεί μια απόφαση ότι το outsourcing των εργών, η ανάθεση δηλαδή σε τρίτους, ε, θεωρούνταν ε, κακή πρακτική. Αυτό έγινε στο πλαίσιο της ε, μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σταδιακά ανακαλύπτουμε και πάλι ότι όταν έχουμε την πρωτοβουλία για καινοτόμες ιδέες θα πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα εκκίνησης μικρότερων έργων με απλούστερους μηχανισμούς και κανόνες που θα μας επιτρέπουν να το πράττουμε αυτό. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Εάν δούμε δηλαδή πώς λειτουργούμε στην πράξη σε ό,τι αφορά την εκτέλεση μικρών τέτοιων έργων Μιλάμε για ένα πραγματικά δυσανάλογο φόρτο διοικητικής εργασίας προκειμένου να τρέξουν τέτοιου είδου έργα. Δηλαδή έχουμε κανόνες οι οποίοι καθοδηγούν αν θέλετε τις ε, μεγάλες δαπάνες σε μεγάλα προγράμματα αλλά και στα μικρότερα έργα. Είμαστε, απαιτείται από εμά να ακολουθούμε τους ίδιους κανόνες για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα 250.000 ευρώ για την διευκρίνηση του πώς θα συνεχιστούν τα έργα σε σχέση με το Erasmus αποτελούν μια καλή δαπάνη, μια χρήσιμη δαπάνη. Δεν θεωρούμε πως χάσαμε χρόνο γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία εξετάστηκαν Αλλά η, η ανάθεση τέτοιων μικρότερων έργων στην, ε, στην ECPRM ε, θεωρήθηκε πως στο παρελθόν τουλάχιστον πως δεν αποτελεί ε, τον ενδεδειγμένο τρόπο εργασίας. Εάν αποφασιστεί στο μέλλον να γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει, αλλά υπό τους τρέχοντες κανόνες, ακόμα και αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να αναθέσουμε δηλαδή σε κάποιον άλλον κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί να υπάρξει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στους ε, παραγωγούς τέτοιων υπηρεσιών με αποτέλεσμα να έχουν δεσμευθεί όλα τα κοντήλια τα οποία θα προβλέπονται για το συγκεκριμένο ε, έργο με αποτέλεσμα όλος ο έλεγχος ή ε, οποιασδήποτε συμπληρωματικές ε, εργασίες που θα πρέπει να γίνουν να αφορούν ήδη αυτό το δεσμευμένο ποσό. Δηλαδή το να προβλέψουμε κάτι συμπληρωματικά δεν θα μας βοηθήσει. Ακόμα δηλαδή και αν πούμε ότι θα υπάρξει μια ανάθεση. Ίσως θα πρέπει ενδεχομένω να εξετάσουμε μια προσέγγιση στο μέλλον σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα του μεγέθους δηλαδή των έργων. Αλλά ε, προς το παρόν, ακόμα και αν έχουμε την καλύτερη τις καλύτερες προθέσεις σήμερα δεν, είναι, πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοί μου θέλουν να κάνουν κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Ε, εν πάση επιτρέψτε μου να αναφέρω και κάτι ακόμα σε σχέση με το Εράσμος. Ε, για να το συνδέσω με κάποια έργα τα οποία δεν τρέχουν. Για παράδειγμα το Ερμπαρτ. Στο Ερμπαρτ Ε, στοχεύουμε κυρίως τις ομάδες εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πελάτες ενός ε, προγράμματος Εράσμους. Οι ανταλλαγές δηλαδή στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΡΜΠΑΤ είναι το να έχουμε α, ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε πολύ συγκεκριμένα ε, project. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ε, λάβουμε κάποιε αποφάσει ό,τι αφορά τα θεματικά παιδιά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν σε τι, ποιο είναι το αντικείμενο στο οποίο εργάζονται και σε σχέση με αυτό συνεργάζονται. Άρα λοιπόν αυτή η ανταλλαγή μέσω του Urbank θα μπορούσε να ε, βοηθήσει ό,τι αφορά την εμβάθυνση αυτή τη ε, προσέγγιση, τη κοινή αντίληψη, τη κοινή κατανόηση, οι οποίοι δρούν με έναν υπεύθυνο τρόπο στον τομέα τη αρμοδιότητα, να εφαρμοστεί. Και να γίνει κάτι τέτοιο είναι εύκολο. Εάν αρχίσουμε να αποσυνδέουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα από κάποιες πιο πρακτικές αν θέλετε εφαρμογές θα μέναμε σε ένα πιο επιφανειακό επίπεδο. Εάν θελήσει κάποιος να πάει πιο βαθιά θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει μια καθοδήγηση και να δώσει να υπάρχει κάποιος συντονιστής, αν θέλετε, ο οποίος ε, θα παρέχει ακριβώς αυτά τα στοιχεία για τον συντονισμό. Δεν νομίζω λοιπόν πως ε, μια πλήρως αν θέλετε αποκεντρωμένη προσέγγιση θα σας ε, απέφερε τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμείτε να δείτε. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλοι συνάδελφοι σας να ζητούν το λόγο. Ε, δυστυχώς είναι συναρμόδιο και ζητήματα απλούστευσης. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να εκφράσουμε εμείς ε, την δική μας επιθυμία για περαιτέρω απλούστευση της ε, πολιτικής εδώ και λύσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την υλοποίηση πιλωτικών projects. Δεν νομίζω πως υπάρχουν άλλα ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Είχαμε καλύψει τα υπόλοιπα, άρα αυτό ήταν το τελευταίο Σήμερα στην διάταξή μας. Σας ευχαριστώ όλου ε, πολύ. Θα σα δω στι στι αρχές Ιουνίου.